όλες οι πολιτικές ομάδες. Υπάρχουν αντιρρήσει. Κάποια πολιτική ομάδα έχει αντίρρηση ω προ το θέμα αυτό, γιατί χρειάζεται πολιτική συμφωνία προκειμένου να κατευθεί μια αναθεωρημένη έκδοση χωρί τι τις αιτιολογικέ σκέψει. Κυρία Βίξτρον, εκ μέρου τη ομάδα μου θέλω και εγώ να συμφωνήσω στα όσα προτάθηκαν. Καθιστώντα όμω σαφέ το εξή με ένα σχόλιο, ότι όταν υπάρχει συμφωνία για το μέλλον, το να ξανανοίγει θέμα στο οποίο έχουμε συμφωνήσει, γιατί δεν θέλω αυτό να αποτελέσει προηγούμενο, Πρέπει να είμαστε λοιπόν σαφείς ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια δυνατότητα να ξανανοίγουν θέματα. Έχουμε δουλέψει για χρόνια στο θέμα αυτό και την ίστατη ώρα, την ώρα που έχει ολοκληρωθεί το κείμενο, βλέπουμε αυτές τις αλλαγές. Λοιπόν, ε, δεν αποτελεί καλό προηγούμενο και παράδειγμα για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία και να μην ξανανοίγουν, να τηρούνται οι συμφωνίες και να μην ε, ανοίγουν πάλι θέματα. Ακριβώς αυτό λέει ο Πρόεδρος. Γι' αυτό και εγώ παρουσιάζοντάς το εξέφρασα τις προσωπικές μου επιφυλάξεις και αντιρρήσει. Είναι ένα σημαντικό θέμα βεβαίως και αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι πια έχει ε, δώσει τέρμα σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις, τις τόσο εντατικές κτλ. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να αποτελέσει προηγούμενο και άκουσα μεν την ε, πρόταση της Επιτροπής. Ο κύριος Έγγελ όμως μάλλον θέλει και αυτό το λόγο. Όχι. Κύριε Κέλλερ, εσά σας είδα σίγουρα. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Βουίσκστρομ ότι ναι, στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχουμε αντιρρήσεις, αλλά επί της αρχής οπωσδήποτε και ίσως θα έπρεπε να συνοδευτεί αυτή η τροποποίηση με μια γενική δήλωση ότι δεν θέλουμε να επαναληφθεί στο μέλλον. Καλώς, εφόσον γίνεται αντιληπτό αυτό, μπορούμε να υποβάλουμε για την Ολομέλεια αναθεωρημένο κείμενο που θα υπογράψω εγώ για να ξανακαταθέσουμε με βάση την πολιτική συμφωνία στην οποία προφανώς καταλήξαμε Κύριε Γκύο. Κύριε Πρόεδρε, με ταυτόχρονη έκφραση βαθιά δυσαρέσκεια ω προ την τροποποίηση που μα προτείνεται την ίστατη ώρα, την ώρα που πρόκειται να ψηφίσουμε ουσιαστικά, μας λέτε ότι μπορεί να προκύψει μια πολιτική συμφωνία και το δεχόμαστε μεν, αλλά ε, ε, υπογραμμίζω και επιμένω στο γεγονός ότι χρόνια, και αναφέρθηκε αυτό, χρόνια τώρα δουλεύουμε το θέμα αυτό, με περίπλοκες συζητήσεις, με αδιέξοδα και διεξόδους και νομίζω ότι τέτοιου είδους μέθοδοι της τελευταίας στιγμής είναι πολύ δύσκολο να γίνουν παραδεκτές ε, ας το δεχθούμε τώρα, αλλά δεν θέλουμε και το κάνουμε για να μην υπάρξει αποσταθεροποίηση στο θέμα αυτό που όπως είπα απέτησε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις επώδυνες πολλές φορές μερικές, ε, πολλές φορές μάλιστα, αλλά δεν θέλουμε να το ξαναδούμε αυτό μπροστά μας. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, πολιτική συμφωνία λοιπόν και παρουσιάζουμε την τροπολογία στην Ολομέλεια της προσεχούς εβδομάδας. Και σας ευχαριστούμε κύριε Κιακαϊόλα. Ψηφοφορία λοιπόν. Κύριε Έγγελ. Κύριε Πρόεδρε και σύντομα για να μην σας καθυστερώ. Από ό,τι φαίνεται και οι συντονιστές συζήτησαν το θέμα της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα. Έκθεση όμως δεν έχουμε ακόμα. και φαίνεται ότι θα γίνει η παρουσίαση στην προσεχή συνεδρία τη Επιτροπής μας. Εγώ ως μέλος αντιπροσωπεία θέλω πριν από τη συζήτηση να δω τη γραπτή έκθεση. Γι' αυτό παρακαλώ, εάν δεν υπάρχει έκθεση για την αποστολή, να αναβληθεί και πάλι η συζήτηση. Τελευταία ανάλυση από το Σεπτέμβριο την έχουμε κάνει. Εάν δεν την συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρία, τη συνεχίσουμε στη μεταπροσεχή. Αλλά να έχουμε την έκθεση πριν. Καλώς λέει ο Πρόεδρος βεβαίως και γι' αυτό ακριβώς καθυστερήσαμε μερικά λεπτά γιατί θέλαμε να κλείσουμε το θέμα αυτό στην συζήτηση των συντονιστών, ήταν το τελευταίο. Μας απασχόλησε για κάμποση ώρα. Θα κυκλοφορήσει αρχές προσεχούς εβδομάδας η έκθεση. Ίσως και αύριο ακόμη λέει η γραμματεία. Η οποία δεσμεύεται αύριο να σας καταθέσει τα πρακτικά της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα. Το σημειώνουμε λοιπόν. Το ταχύτερο δυνατό θα γίνει. Και τώρα προχωράμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε αυτά τα θέματα και μάλιστα εγκαίρως. Έχουμε το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Επιθέσεις κατά πληροφορικών συστημάτων απόφαση του Συμβουλίου. Κυρία Χολμάιερ είναι η συγκεκριά και υπενθυμίζω ότι πρόκειται για ένα από τα θέματα που μας έχουν απασχολήσει σχετίζονται με τη διαδικασία του Σέγγεν, το έχουμε υπόψη και τώρα συνεχίζουμε στη διαδικασία αυτή που μας φέρνει αντιμέτωπο με μια πρώτη ψηφοφορία. Σα θυμίζω ότι χρειάζεται η ηλεκτρονική σας κάρτα και αν έχετε τον κατάλογο των ψηφοφοριών μπορούμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. First. Πρώτα πρώτα, το συμβαστικό κείμενο. Τροπολογία υπαριθμών 129. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία. Που σημαίνει ότι πάμε κατευθείαν στη σελίδα υπαριθμών 9 του καταλόγου της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Now the vote is closed. Πέρα ψηφοφορίας. 36 υπέρ 8 κατά. Καμία εποχή, επομένως εγκρίνεται. Και ευχαριστούμε την κυρία Μόνικα Χολ Μάιερ για την έκθεσή της. Και τώρα έχουμε την επομένη έκθεση. Η τροπολογία όσον αυτό αφορά την ε, Συμφωνία Σέγγεν. Η συγκριτής είναι ο κ. παπα Θέλετε το λόγο? Όχι. Να ευχαριστήσω του και ηγητέ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τη Γραμματεία μα. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και κατά τι διαπραγματεύσει. Και προχωρούμε στην ψηφορία, λέει ο Πρόεδρο. Ο εισηγητή προτείνει να ψηφίσουμε μαζί όλε τι διατάξει για την τροπολογία 82 σαν συμβαστικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά αποχές επομένως εγκρίνεται το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε κατευθείαν στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά Now the vote is closed. Ψηφίζουμε πέρα της ψηφοφορίας. 41 υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή. Ευχαριστούμε τον κύριο και τώρα πηγαίνουμε στα σημεία που θα συζητηθούν. Στο σημείο υπαριθμών 6 και το 7 θα συζητηθούν από κοινού. Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρασίνου Ακροτηρίου όσον αφορά την επανεισδοχή ε, προσώπων που παρανόμως διαμένουν στη χώρα. Η συγκεκριμένη είναι η κυρία Μαρία Γκαμπριέλ και το σημείο υπαριθμών 7 που αφορά τη συμφωνία μεταξύ πάλι Ευρωπαϊκή Ένωση και Πρασίνου Ακροτήριου όσον αφορά την διευκόλυνση για κάποιε θεωρήσει διαβατηρίων ε, μικρή διάρκεια. Θα πρέπει να συζητήσουμε τα σχέδια κειμένου για αυτές τις δύο εκθέσεις. Και δίνουμε το λόγο στην συγκίτρια την κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα πρώτα. Αρχίζω τονίζοντας πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δύο εκθέσεις. Διότι για πρώτη φορά πρόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσουμε για αυτή τη συμφωνία μεταξύ ε, μιας ε, χώρας της Αφρικής και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Αφρική και είναι πάρα πολύ σημαντική. Επομένω, η σύνοψη αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρασίνου Αγροτηρίου. Να σα ξεκινήσουμε πρώτα πρώτα με το ιστορικό για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας Πρασίνου Αγροτηρίου. Πρώτα πρώτα έχουμε συμφωνία Κοτονού μεταξύ ΑΚΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχει και εταιρική σχέση για την ε, κινητικότητα ε, των προσώπων μεταξύ των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί στα πλαίσια της πολιτικής πέραν των ε, παραδοσιακών ε, σχέσεων και ο στόχος είναι να εμβαθύνει τις σχέσεις με τη δημοκρατία του Πρασίνου Ακροτηρίου, ούτω ώστε να υπάρχει ε, καλή διακυβέρνηση, σταθερότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και καταπολέμηση της φτώχειας. Επίσης, να ληφθεί υπόψη η κοινωνία της κατάρτισης, της γνώσης και τα πολιτιστικά. Είναι μια δημοκρατία σταθερή όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σεβαστά εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε μια ανακοίνωση όσον αφορά τι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας αυτής. Σε αυτή την ανακοίνωση η Επιτροπή αναγνώρισε ότι υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των δύο μερών. Και ε, επίσης ε, ότι υπάρχουν κοινέ κοινωνικοπολιτικές αξίες. Το υψηλό επίπεδο των προτύπων και πρακτικών της χώρας αυτής για τη διακυβέρνηση ε, αποτελεί βάσιμο λόγο για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία για εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρασίνου Ακροτηρίου είναι κάτι το οποίο θα συμβάλλει σίγουρα στη βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης και στο σεβασμό των ελευθεριών. Έχουμε επομένω αυτές τις δύο συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη διευκόλυνση θεωρήσεων βραχίας διαμονή. Η δεύτερη συμφωνία αφορά την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. Ως εισηγήτριο. Εγκρίνω τη σύναψη αυτών των δύο αλληλοεξαρτωμένων και παραλλήλων συμφωνιών. Πρέπει ταυτόχρονα να τεθούν σε ισχύ. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τώρα ευρύτερα όρια για ελευθερία, ασφαλή και δικαιοσύνη. Και πέραν τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, αυτέ οι δύο συμφωνίε καταρχήν αποτελούν ένα σημαντικό βήμα. Εξέλιξη για τις σχέσεις Ένωσης και Πρασινού Ακροτηρίου. Και επομένω, πέραν της σύναψη της συμφωνίας ε, υπάρχει ε, ιδιότητα βαρύνουσα σημασία. Επίσης, θα τονίζω ότι αυτές οι συμφωνίες προσφέρουν ενδιαφέρον σε περιφερειακό επίπεδο. Θα συμβάλλουν στις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναβάθμιση συνεργασίας και με άλλες χώρες εκεί. Για το πράσινο κρατήριο βεβαίως αυτό είναι πρόοδος, ενθάρρυνση για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε τώρα τι γίνεται για αυτές τις ε, συμφωνίες. Πρώτα πρώτα, η πρώτη που αφορά την έκδοση θεωρήσεων βραχίας διαμονή. Αυτό θα γίνει με αμοιβιότητα. Η έκδοση θεωρήσεων για τους πολίτες Πράσινου και της για διαμονή που δεν θα είναι πάνω από 90 μέρες σε περίοδο 180 ημερών. Επίσης, θα έχουμε απλουστευμένες προϋποθέσεις για θεωρήσεις πολλαπλές. ισχύω 5 ετών. Παραδείγματος χάρη για μελικυβερνήσεων, ε, μέλη αντιπροσωπιών με διάρκεια δύο ετών που θα καλύπτει δημοσιογράφους, φοιτητές κλπ. Πολλαπλές εισόδους επίσης ε, προβλέπουν κάποιες θεωρήσεις για δύο έτη, πέντε έτη όταν έχουμε κάποιον που έχει ζητήσει τη θεώρηση και έκανε καλή χρήση της θεώρησης και όταν η πρόθεση των ταξιδιών δεν αφορά περιορισμένο διάστημα. Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από τις θεωρήσεις για μέλη αντιπροσωπιών, για παιδιά κάτω των 12, μαθητές, φοιτητές, νέους έως 25, για σεμινάρια και επίσης ε, θα προβλέπεται και 30 ευρώ ως έξοδα για την θεώρηση. Ε, παράταση επίσης προβλέπεται για αυτούς που δεν μπορούν να βγουν από το έδαφος κατώμενο προς ε, ε, για λόγους ανωτέρας βίας. Επίσης, περιορισμένη απαλλαγή για υπηκός προς ακροτηρίο που έχουν πλαντικό διαβατήριο ή υπηρεσιακό και για αυτούς οι οποίοι έχασαν ή τους έκλεψαν κατά την παραμονή τους τα, Επίσης έχουμε την συμφωνία για την επανεισδοχή και εδώ με αμοιβαίο τρόπο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και αφορά επίσης τους πάτριδες και τους ε, πολίτες των χωρών. Καλύπτονται επίσης τα μέλη της οικογένειας τους, σύζυγος και ε, ανήλικα παιδιά και, και υπάρχουν επίση και κάποιες ε, άλλες ε, τεχνικές προϋποθέσεις που καθορίζονται και θα πρέπει βεβαίως να αποδεικνύεται η ηθαγένεια. Αυτή η, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές μέσα σε δύο εργάσιμες μέρες. Ε, μπορεί να έχουμε και μια ταχεία διαδικασία προβλέπεται και η φυσιολογική διαδικασία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η συμφωνία για την επανεισδοχή επίσης περιέχει και κάποιες διατάξεις όσον αφορά την διαμετακόμιση ή το, transit και, υπάρχει αντιστοιχεία με τις δεσμεύσεις από τις διεθνείς συνθήκες που για να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις δύο αυτές ε, συνθήκε, λαμβάνει υπόψη το τι ισχύει για Δανία, Ενωμένο Βασίλειο ε, και Ιρλανδία και στις, ε, υπάρχουν κάποιε κοινέ ε, δηλώσει που επισυνάπτονται, αλλά και στην αιτιολογική έκδοση. Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία και εκεί επίση υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσει σε σχέση με, το, με, το, με, με την περιοχή του Σέγγεν και υπάρχει τέτοια σχετική κοινή δήλωση. Πρώτα-πρώτα, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλοκεί όσον αφορά την έναρξη και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ε, για τι συμφωνίε τέτοιου είδου. Συνιστώ επίση το Κοινοβούλιο να εποπτεύει την εφαρμογή των συμφωνιών. Επίση, να μπορεί να συμμετάσχει στο, στη, στη δομή που υπάρχει για την εφαρμογή, δηλαδή στην μεικτή διαχειριστική επιτροπή. Άρα, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει κάποια στιγμή αυτές τις μεικτές επιτροπές για τη διαχείριση των συμφωνιών. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σε όλες τις φάσεις για την εφαρμογή των συμφωνιών σύμφωνα με την αρχή καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Με μια φράση που όμως συμπεράσματος, θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη της Επιτροπής μα να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή. Ο πρόεδρο! σας ευχαριστούμε εμείς, κυρία Μαρία Γκαμπριέλ. Και τώρα το λόγο έχουν οι σκιώδει Κύριε Αντανούκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μας έχουμε αυτή την ε, δέσμη του συμπίνου αυτών των δύο συμφωνιών. Η πρώτη όσον αφορά τις θεωρίες διαβατήριων και η άλλη όσον αφορά την επανεισδοχή. Βάλετε ταυτοχρόνως να διεκπαιρεώσουμε αυτές τις ε, δύο συστάσεις. Εμείς πάντως είμαστε κατά μιας δύο προσέγγισης. σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε κατά τη ε, συμφωνία επανεισδοχή. Σα υπενθυμίζω, δε, ε, ότι το πράσινο ακροτήριο δεν είναι χώρα που έχει προσυπογράψει την ε, συμφωνία του ΟΗΕ για το καθεστώς που διέπει τους πρόσφυγες. Άρα δεν είναι σωστό εμείς, αφού είμαστε ένα όργανο δημοκρατικό, να υποστηρίζουν μια τέτοια συμφωνία επανεισδοχής με τη χώρα εκείνη. Βεβαίω και είμαστε υπέρ τη ε, συμφωνία για πλούστευση εκδόση θεωρήσεων, αλλά όχι για την επανεισδοχή. Βεβαίω και πρέπει να συγχαρούμε παρά τη διαφωνία μας την εισηγήτρια για το έργο επιτέλεση. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω τώρα μήπω ε, η Προεδρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Well, thank you, Mr. Chairman. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις συμφωνίες όσον αφορά την κύρωση αυτών των ε, δύο συμφωνιών που αποτελούν ε, ενία δεσμημέτρων. Όταν τεθούν σε ισχύ αυτές οι δύο συμφωνίες θα έχουμε κάνει ένα βήμα πρώτο παραπάνω σε σχέση με την προσέγγιση ε, Πρασινοκροτηρίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα έχουμε καλύτερη κινητικότητα προσώπων, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μόνο μία παρατήρηση προς την ε, εισηγήτρια όσον αφορά την ε, ε, σύνθεση των, της μεκτής Επιτροπής. Βεβαίως και θα το κοιτάξουμε. Αλλά βέβαια θα πρέπει να μην ξεχνούμε ποτέ τη θεσμική ισορροπία. Σαφές είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι κι αλλιώς θα εμπλακεί στην εποπτεία για την εφαρμογή των συμφωνιών, θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο. Επομένως αυτό ήδη έχει ληφθεί υπόψη και έχει αναλάβει τις σχετικές συνέργειες η Γενική μας Διεύθυνση. Επίσης, με την νομική μας υπηρεσία θα εξετάσουμε κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμμετάσχει στις εργασίες της Μικτής Επιτροπής για ε, αυτές τις ε, συμφωνίες, ιδίως όσον αφορά τις θεωρήσεις. λάβουμε επίσης υπόψη τι είπε η σκιώδη συγκεντρία. Ο Πρόεδρος, ολοκληρώσατε. Um, Κάτι για την επανεισδοχή να προσθέσω. Δύο σύντομα σημεία. Πρώτα πρώτα τη σχέση μεταξύ διευκόλυνση θεωρήσεων και επανεισδοχής. Βεβαίω. Και εδώ είναι θέμα επιλογή και θέμα επιλογή του Πασίνου Πετρίου, αλλά εγώ θα θέλω να σα τονίσω το ότι η διευκόλυνση για τι θεωρήσει ε, θα, θα εξαρτηθεί για το πότε θα ισχύσει από την άλλη συμφωνία. Εάν επομένως σε μία συμφωνία δεν κυρωθεί, τότε σαν συνέπεια θα ανασταλεί και η θέση σε ισχύ τη άλλη συμφωνία. Αν δεν έχουμε πρώτη την επανεισδοχή δεν θα έχουμε ούτε τι θεωρήσει και τη διευκόλυνση. Τώρα όσον αφορά την ε, Συμφωνία της Γενέβης, ε, στο πρωτόκολλο 67 έχει προσχωρήσει το πράσινο κριτήριο και επίσης στην άλλη συμφωνία το 87. Έτσι κι αλλιώς ε, αυτή η συμφωνία πανεισδοχής δεν μπορεί να, να, να ακυρώσει τις δεσμεύσεις οποιοδήποτε των μερών από διεθνείς συμφωνίες. Το Συμβούλιο έχει κάποια παρατήρηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι πολύ σύντομο και απλώ θα ήθελα να σα πω από πλευρά τη Προεδρία και του Συμβουλίου ότι θεωρούμε πολύ θετικέ αυτέ τι συμφωνίε και συμφωνούμε με όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι σημαντικό αυτά να τα διεκπαιρώσουμε μαζί σαν δέσμη μέτρων. Οπότε θα πρέπει και αυτά να προωθηθούν από κοινού δύο συμφωνίες. Πολύ σημαντικά αυτά και για τις χώρες ΑΚΕ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που μια χώρα ΑΚΕ συνήψε τέτοια συμφωνία. Επομένω θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και είμαστε υπέρ. Κύριε Γκαμπρίελ, θέλετε εσείς να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σντανόκα και την Επιτροπή και το Συμβούλιο για όσα είπαν Επίσης, Πρόεδρε, θα ήθελα να μας πείτε τι προβλέπετε σαν προθεσμοί για τις τροπολογίες κλπ. Να διευγανιστεί αυτό, τόσο ώστε να ξέρουν οι συνάδελφοι τι θα γίνει με τις τροπολογίες που θέλουν τυχόν να καταθέσουν. Τι προθεσμία θα καθοριστεί. Βεβαίω, βέβαια, λέει ο Πρόεδρος, θα σας πω. Προθεσμία για τις τροπολογίες 13 Μόνο διαδικαστικού χαρακτήρα τροπολογίες θα είναι παραδεκτές. Και 8 ή 9 Ιουλίου θα κάνουμε την ψηφορία. Άρα, γιατί υπόψη αυτή θα είναι η 9 ιουλιου θα κανουμε την ψηφορια αρα για την υποψη αυτη θα ειναι η προθεσμια 13 Ιουνίου για διαδικαστικού χαρακτήρα τροπολογίες. Καλώς, ωραία και σας ευχαριστούμε που έχετε συμμετάσχει στη συζήτηση αυτή για το πράσινο κρατήριο για αυτές τις δύο συμφωνίες. Την εποπτεία των εξωτερικών ε, θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Frontex και τα κράτη-μέλη. Έχουμε τον εισηγητή μας συνάδελφο Κάρλος Κοέλιο και θα πρέπει να έχουμε υπόψη πως αυτό το θέμα έχει συζητηθεί πριν από χρόνια όταν η Κομισιόν πρότεινε τις κατευθύντες γραμμές για την εποπτεία των θαλασσίων συνόρων υπό την επιτροπολογία, αλλά θεωρήθηκε ότι ήταν εκτός ε, των ε, αρμοδιοτήτων της ε, επιτροπολογίας. Οπότε το θέμα ήρθε ενώπιον του ΔΕΚ και η Κομισιόν κέρδισε και έκανε και πρόταση υπό την φυσιολογική νομοθετική διαδικασία και θα ακούσουμε μια έκθεση τις πρώτες δηλαδή παρατηρήσεις του κυρίου Κοέλιο και μετά θα συζητήσουμε. Παρακαλώ κύριε Κοέλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως μόλις είπατε, το θέμα αυτό ξεκινά επί τη βάση μιας νομικής νίκης του Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας δικαίωσε και ακύρωσε την απόφαση που είχε ληφθεί από το Συμβούλιο και η πρόταση που υποβάλλει τώρα η Κομισιόν αντικαθιστά την απόφαση του Συμβουλίου. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης πως οι επιπτώσεις της, αποφάσης, της αυτής θα διατηρηθούν μέχρι ότου να υπάρξει ένας κανονισμός που να υποκαθιστά αυτήν την κατάσταση. Και το επίσης διευκρινίζει ότι θα πρέπει να γίνει αυτό σε κάποιο λογικό χρονικό πλαίσιο. Δεν ορίζει τι είναι κάποιο λογικό πλαίσιο, αλλά θα πρέπει αυτό να λειτουργήσει ως κίνητρο ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτό το θέμα, ούτως ώστε ο κανονισμό μας να μπορέσει όσο γίνεται πιο σύντομα να αντικαταστήσει την απόφαση που έχει ακυρωθεί και που εξακολουθεί να ισχύει. Πάντως υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά την ερμηνεία του Διεθνούς Θαλασσίου Δικαίου και τις ε, ισχύουσες πρακτικές. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ε, νομική αβεβαιότητα, μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα επιχειρήσεων που συντονίζονται από τη Frontex, μπορεί επίσης να αιτιολογήσει μια ισχνή συμμετοχή των κρατών μελών, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, υλικό, πόρους ανθρώπινους και βεβαίως αυτό μπορεί να, θέσει, να αμφισβητήσει την αλληλεγγύη που είναι τόσο απαραίτητη για την σωστή υποπτία των εξωτερικών μας ε, ε, θαλασσίων συνόρων. Γι' αυτό και συμφωνούμε ε, ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινοί κανόνες για την εποπτεία των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων μας στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που τη συντονίζει η Frontex. Και θα ήθελα να πω ότι η Frontex με τη διάρκεια των ετών τελικά δίνει μια πολύτιμη βοήθεια στα κρατη Αν λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκε στη τελευταία έκθεση για το Σέγγεν, το έκθεση που μας παρουσίασε η Κομισιόν στα τέλη του περασμένου μήνα, είναι ε, ε, ξεκάθαρο ότι έχουν υπάρξει σημαντικές πρόοδοι. Τώρα, επί της ουσίας της πρότασης της Κομισιόν, εγώ θα πρέπει να πω ότι μου φαίνεται αρκετά ισορροπημένη γιατί ενσωματώνει ε, ε, ένα κομμάτι των μέτρων που ήδη υπήρχαν διατηρεί διάφορες επιχειρήσεις, δηλαδή την εποπτεία που κάνουν τα κράτη-μέλη με το, υπό τον συντονισμό της Frontex αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξής. Καταρχήν υπάρχει εγγύηση μιας αποτελεσματικής εποπτείας τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η διέλευση η μη ε, εγκεκριμένη και ε, να καταπολεμηθεί η συνοριακή εγκληματικότητα. Η πρόταση διευκρινίζει επίσης την ε, έννοια της εποπτείας των συνόρων. Δεν καλύπτει απλώς τη διέλευση την άτυπη προέλευση, την ατυπική αντικανονική διέλευση, αλλά ορίζει μέτρα ε, εντοπισμού αναζήτησης έρευνας ε, σύμφωνα με τους διεθνείς ισχύοντες κανόνες για να μπορέσει να βοηθήσει άτομα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου. Και ο κανονισμός είναι πληρέστερος όσον και ακριβέστερος όσον αφορά την προστασία των ε, βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Από τη στιγμή που δούμε λοιπόν τα μέτρα, διευρύνονται έτσι τα μέτρα για την ε, διάσωση και την ε, έρευνα. Γίνεται δηλαδή μια απόπειρα για να δημιουργηθεί ένα σύνολο μέτρων εγγυήσεων ουσιαστικών έτσι ώστε να είναι βέβαιο πως ε, κατά την αποβίβαση ανθρώπων που λαθρέα έχουν περάσει τα σύνορα να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατόπιν τούτων όλων θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ε, ε, θα πρέπει να εργαστούμε με επιταχυμένο τρόπο, να μην πω βέβαια υπό κατεπίγουσες συνθήκες, αλλά γρήγορα, ώστε να εγκριθεί γρήγορα ο κανονισμός που θα πρέπει να αντικαταστήσει την απόφαση, η οποία εντωμεταξύ στη μεταβατική περίοδο εξακολουθεί να ισχύει. Εγώ από πλευρά μου συζητήσει είμαι διαθέσιμο, να προσπαθήσουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να βρούμε συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Θα ήθελα να ζητήσω τη συνεργασία των σκιωδών εισηγητών έτσι ώστε αυτό το σφιχτό χρονοδιάγραμμα να τηρηθεί γιατί θα επέτρεπε όπως σας είπα να αντικατασταθεί η απόφαση. Έχω την φοβούμε πως αν δεν τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος του έτους, με, καθώς θα πλησιάζει η εκλογική περίοδος για το Ευρωκοινοβούλιο, δεν θα καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέσα στη διάρκεια αυτής της θητείας και θα αναβληθεί για το 2015, ενώ η απόφαση αυτή έχει ήδη ακυρωθεί από το δικαστήριο. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε κύριο Κοέλιο. Να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Κομισιόν που μόλις κατέφτασε. Πείτε μας τη γνώμη σας γιατί θα θέλαμε ο εισηγητή μας να μας κάνει μια, ένα σχέδιο έκθεσης ε, μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Γι' αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε πού βρίσκεται το θέμα από την προοπτική της Κομισιόν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, εμείς έχουμε προσπαθήσει να κινηθούμε όσο γινόταν πιο γρήγορα. Υποβάλαμε την πρόταση αυτή μετά από την απόφαση του ε, δικαστηρίου είχαμε επαφές με βουλευτές αλλά και με τη Frontex για να λάβουμε υπόψη τις εμπειρίες που ε, έχει αποκομίσει μετά από την εφαρμογή της απόφασης αυτής και επίσης τη γνώμη τους για τις, ε, τις ουσίες αλλαγές στη νέα πρόταση στην ουσία επιδιώκει τους ίδιους στόχους όπως και η ακυρωμένη απόφαση ε, πρέπει, θέλει να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων της Frontex στα ευθαλάσσια σύνορα, να ενθαρρύνει την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή κρατών μελών σε αυτές τις επιχειρήσεις σε πνεύμα αλληλεγγύης και τέλος να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και να δημιουργήσει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για αυτές τις επιχειρήσεις. Οι στόχοι λοιπόν παραμένουν οι ίδιοι βασικά, είναι οι ίδιοι και με τη νέα πρόταση με την έννοια ότι εστιάζουμε στον συντονισμό των επιχειρήσεων από τη Frontex στα θαλάσσια σύνορα. Η μορφή βέβαια αλλάζει, οπότε τώρα είναι πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ένα, μια σημαντική διαφορά επί της μορφής, ωστόσο σε σύγκριση με την απόφαση είναι ότι η παλαιά απόφαση του Συμβουλίου είχε χωριστεί σε δύο κομμάτια, ένα δεσμευτικό και ένα μη δεσμευτικό, ενώ τώρα προτείνεται όλοι οι κανόνες και ο κανονισμός εν γέννη να είναι απόλυτα δεσμευτικοί ε, Επί της ουσίας τώρα, χωρίς να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες τώρα, νομίζω πως κάποια στοιχεία θα σας δείξουν ότι έχουμε αναπτύξει περισσότερο ε, την αρχή του non refoulement να λαφθεί υπόψη σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απόφαση Hirsing όπως αποκαλείται, Επίσης και εδώ ε, για να είμαστε βέβαιοι πως θα υπάρχει κοινή συνεννόηση για τα κράτη-μέλη για το πώς στην πράξη θα εφαρμόζουν αυτή την αρχή. Επίσης έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε λεπτομέρειες για τις επιχειρήσεις έρευνας, αναζήτησης και διάσωσης, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον διεθνές δίκαιο, καθώς και λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη αυτές οι αρχές ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οποιοδήποτε χρειάζεται διάσωση θα διασωθεί και ότι τα κράτη-μέλη θα λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων Frontex. Και τελευταίο σημείο επί της ουσίας είναι ότι αναθεωρήσαμε κάπως τους κανόνες για την αποβίβαση, ώστε να είμαστε βέβαιοι και πάλι ότι σεβαγόμαστε το ισχύον διεθνές δίκαιο, να υπάρχει ευελιξία αλλά και να υπάρχει και σαφής υποχρέωση των κρατών μελών να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά και με στο κέντρο συντονισμού της διάσωσης για να μπορούν να αποβιβαστούν οποιοδήποτε μετανάστες έχουν συλλεχθεί στη θάλασσα και να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλειά τους. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι, ότι καλωσορίζω τη δέσμευση του εισηγητή να κινηθούμε γρήγορα και εμείς το ίδιο μήνυμα στείλαμε στο Συμβούλιο ότι ελπίζουμε να θεωρηθεί προτεραιότητα το θέμα αυτό ώστε να είμαστε βέβαιοι πως θα έχουμε το νέο μέσο στην διάθεσή μας ώστε να αντικατασταθεί η απόφαση του Συμβουλίου για στόχους νομικής βεβαιότητας και σαφήνειας. Σας ευχαριστώ. Την Κομισιόν η, η Προεδρία έχει να σχολιάσει κύριε Ντουάιερ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ με το όσο είπε ο ότι ε, δηλαδή θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα η εργασία μας πάνω σε αυτό το ντοσιέ, γιατί είναι ένα μέτρο προτεραιότητας για το Συμβούλιο και ε, ότι θα πρέπει αυτό να ε, το επεξεργαστούμε σε ένα λογικό χρονικό διάστημα είναι στο μυαλό μας. Η Κομισιόν υπογράμμισε ποιο είναι το περιεχόμενο και λεπτομέρειε της πρότασης. Ε, τώρα όσον αφορά τη διαδικασία, το θέμα υποβλήθηκε στην ΣΚΙΦΑ. Η ΣΚΙΦΑ κάλεσε την ομάδα εργασίας για τα σύνορα να εξετάσει τις λεπτομέρειες του ντοσιέ και τώρα αυτή η δουλειά θα ξεκινήσει. Όπως σας είπα, είναι προτεραιότητα. Το λέω γνωρίζοντα το γεγονό ότι η Ιρλανδική Προεδρία σύντομα θα ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Λιθουανοί συνάδελφοι που θα αναλάβουν από τον Ιούλιο θα το θεωρήσουν και εκείνοι προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Έλερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον εισηγητή. Βεβαίως είμαστε πρόθυμοι να να, να συμβάλλουμε και εμείς ώστε να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα ε, η εξέταση αυτού του θέματος. Ευχαριστούμε την Κομισιόν που το έχει θέσει επιτάπητος. Έχω όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ναι, Αν δούμε τη σελίδα 5... όπου μιλάει για το περιεχόμενο και όπου λέτε ότι Ο κόσμος θα πρέπει να ενημερώνεται για το χώρο αποβίβασης και θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να πούν γιατί μπορεί να πιστεύουν ότι αυτό ο χώρος αποβίβασης μπορεί να σημαίνει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Πάντως θέλω να ξέρω τι θα γίνει αν έχουν αντίρρηση να αποβιβαστούν εκεί. Θα πρέπει να τους ρωτήσετε, αλλά τι γίνεται αν όντω εκφράσουν αντίρρηση. Έπειτα, Άρθρο 4 παράγραφος 3 βασικά πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Ε, θα τους δοθεί ευκαιρία να εκφράσουν ε, τους λόγους για τους οποίους και επίσης τι θα πει θα τους δοθεί ευκαιρία. Ευκαιρία μπορεί κάποιος να πει απλώς κάτι ή πρέπει να πας και να τον ρωτήσεις εσύ συγκεκριμένα. Δεν είναι απόλυτα σαφές. Παράγραφος 4 ειδικέ ανάγκες των παιδιών κτλ. Και λήψη υπόψη αυτών, τι θα πει αντρέ όμως που λέτε εδώ, μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα και εδώ θέλω να διευκρινιστεί. Άρθρο 7 παράγραφος 1 C. Τους επιτρέπεται ή δεν τους επιτρέπεται να διανέσουν τα σύνορα. Εκεί δεν είναι ξεκάθαρο και πάλι στο άρθρο 7 Υπάρχει μια διαφορά. Λέει, εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ενώ αλλού λέει βάσιμη υποψία. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο. Article 9, paragraph 9, um, the rescue coordination shall be contacted. Έπειτα λέει ότι Ποιο, ποιο κέντρο διάσωσης και συντονισμού θα έρθουμε σε επαφή. Και τι θα πει έρχομαι σε επαφή. Στέλνω μηνύματα αλλά δεν είμαι βέβαιος τι θα γίνει μετά. Μήπως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως αυτές οι πληροφορίες κάπως κάποιος κάτι της κάνει. Ναι, αυτά είναι οι παρατηρήσεις που είχα να κάνω και στρέφομαι, λέει ο Πρόεδρος, στην Κομισιόν αμέσω ε, για να μας απαντήσει. Είδα και το χέρι της κυρίας Βίκστρομ. Παρακαλώ. Ε, εξ ονόματο τη Άλδη θα πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας κύριε έλιο ε, σε αυτή την έκθεση και καλωσορίζω την πρόταση οι φρικτές ιστορίες που βλέπουμε εδώ και χρόνια και εξακολουθούμε να βλέπουμε κόσμος που θαλασσοπνίγεται στη Μεσόγειο ενώ προσπαθεί να έρθει, φτάσει στην Ευρώπη. Πιστεύω πως είναι ντροπή και αποτυχία όλων μας. Είναι φρικτό και τραγικό να βλέπεις ότι ο κόσμος τόσο απελπισμένος είναι που θέλει να έρθει που μπαίνει σε ένα οποιοδήποτε σκάφος για να φτάσει εδώ. Αλλά ξέρουμε ότι όταν οι ακτοφυλακές των κρατών μελών τα ανακαλύπτουν, αυτά τα καριδότσουφλα δεν κάνουν τίποτα για να σώσουν τις ζωές των ανθρώπων αυτών. Πρέπει πολύ να προσέξουμε την έκθεση του Συμβουλίου των Ευρώπου, την και Στρίκ, είναι υπεύθυνη για τις μάλλον έχει φτιάξει αυτή την έκθεση που ρωτά ποιος είναι υπεύθυνο για τις ζωές που χάνονται στη Μεσόγειο και για τη συγκεκριμένη υπόθεση 62 άτομα χάθηκαν ενώ θα μπορούσαν να έχουν διασταθεί γιατί το ε, μήνυμά τους σημειώθηκε αλλά αγνοήθηκε από αλλιευτικά σκάφη αλλά και από ένα στρατικό ελικόπτερο και ένα στρατιωτικό σκάφος που έπλεε πολύ κοντά εκεί που βρισκόταν το σκάφος που κινδύνευε. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πρόβλημα που Έχουμε διαφορετικούς κανόνες και αντικρουόμενου κανόνες πολλές φορές στα κράτη-μέλη σε σχέση με τι θαλάσσιες επιχειρήσεις. Μα πιστεύω πως σε καταστάσει επίγουσε όταν κινδυνεύουν ζωές θα έπρεπε να είναι δυνατόν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες. Δυστυχώς μέχρι στιγμή αυτό δεν έχει πάντοτε γίνει στην πράξη. Γι' αυτό και ε, θεωρώ ότι είναι κάτι που πραγματικά ε, θα έπρεπε να μας δεσμεύσει να κάνουμε κάτι, να βρούμε λύση. Πρέπει να συντονίσουμε τους κανόνες μας και τις προσπαθίες μας και οι κανόνες να είναι ε, απόλυτα ξεκάθαροι για όλους, να μην υπάρχει καμιά απολύτως αμφιβολία για το ποιος είναι υπεύθυνο και τι πρέπει να κάνει σε τέτοιου είδους περιστάσεις επίγουσες. Όπως συμφωνήθηκε όταν δόθηκε η νέα εντολή στο, στη Frontex, όλες οι δραστηριότητες της υπηρεσίας θα πρέπει να εξεταστούν ε, πολύ προσεκτικά από ε, την άποψη των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτές οι δραστηριότητες ακόμα και να πάψουν αν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. Και θυμάμαι πόσο πολύ που αγωνιστήκαμε για να μπει αυτό στο, κείμενο. Τώρα υπάρχει και θα πρέπει να εφαρμόζεται η υπηρεσία έχει να παίξει ρόλο από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη έχουν φανεί ανίκανα να αναλάβουν την ευθύνη τα ίδια. Η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι ιδιαίτερη ε, και χρειάζεται κοινή, κοινοτική προσέγγιση για να το αντιμετωπίσουμε και να μην αφήσουμε μόνο τα κράτη της περιοχής να το αντιμετωπίσουν. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά θέλω να αναφέρω κάποιες ανησυχίες. Καταρχήν, θα πρέπει να αποσαφινιστεί πως η αρχή του non-refoulement καλύπτει όλους, όχι μόνο πρόσφυγες ή ζητούντες άσυλο. Και επίσης ότι θα γίνεται σεβαστή αυτή η αρχή σε κάθε περίπτωση. Και δεύτερον θα πρέπει να αποσαφινιστεί πως όταν μια μεταφορά δεν μπορεί να γίνει διότι υπάρχει κίνδυνος απάνθρωπης ή αναξιοπρεπούς μεταχείρισης και παραθέτω το νέο άρθρο 3.2 στον νέο κανονισμό του Δουβλίνου επί του οποίου έχω εργαστεί για τόσο πολύ καιρό και που αφορά τρίτες χώρες καθώς και χώρες της Ένωσης ε, σωστή αξιολόγηση των, προστασία, των αναγκών προστασίας των ανθρώπων δεν μπορεί να γίνει πάνω στα σκάφη και η αποβίβαση δεν μπορεί να γίνει εκεί όπου μπορεί οι αποβιβαζόμενοι να ε, αντιμετωπιστούν άσχημα ή να παραβιαστούν τα δικαιώματά τους, τα ανθρώπινα τους δικαιώματα. Ανησυχώ κάπως για τις φήμες τώρα που κυκλοφορούν ότι το Συμβούλιο και η υπερχόμενη ε, Προεδρία δεν έχουν φιλόδοξη ατζέντα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ πραγματικά πιστεύω να είναι απλώς φήμες και τονίζω την ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα για το θέμα. Ελπίζω πραγματικά πως η Λιθουανική Προεδρία και το Συμβούλιο θα ασχοληθούν με το θέμα, θα το ε, δώσουν προτεραιότητα έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι πώς θα προχωρήσουμε προς το συμφέρον όλων μας και προς το συμφέρον της προστασίας της αξιοπιστίας της Ένωσης. Ευχαριστώ. Η Ας δούμε λοιπόν. Τι θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που έθεσαν οι βουλευτές. Ένα από τα θέματα που θα να έχω αναφέρει μάλλον εξ αρχή είναι ότι πρέπει την ερώτηση αυτή να την κοιτάξουμε παράλληλα με τον νέο κανονισμό Frontex και τις εγγυήσεις που βλέπουμε στη νέα τροποποίηση και σε συμπληρώση του κανονισμού είναι συμπληρούμενο αυτά. Στα πιο συγκεκριμένα θέματα και κυρίως στο άρθρο 4 οι στόχοι που θα προσδοριστούν σε σχέση με κάποιον που συλλέγεται στη θάλασσα, από τη θάλασσα ε, είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουν να λάβουν την απόφαση για την τήρηση του, των αρχών αυτών τα κράτη-μέλη. Επίσης, η αναφορά ότι αυτός που περισλέγεται στη θάλασσα ε, θα πρέπει να έχει δικαίωμα σε μια πιο ε, θετική στάση του πληρώματος και όχι απλώς την καταγραφή της κατάστασής του, αλλά φροντίδα. Είναι ένα άλλο θέμα. Είναι δύσκολο βέβαια. Πολλές φορές στη θάλασσα, τα ανοιχτή θάλασσα, υπό δύσκολε συνθήκες, μερικές φορές να επιτελεθεί αυτό το έργο, αλλά εάν δεν είναι δυνατόν να προβεί στην αξιολόγηση αυτή, δεν μπορεί να προχωρήσει σε απόβαση σε τρίτο σκάφος, ώστε να μην παραβιάσει το δίκαιο. Για την παράγραφο τη με τις ειδικές ανάγκες. Είναι δύσκολο να δώσουμε συγκεκριμένα και πρακτικά παραδείγματα. Υπάρχει μια σειρά από καταστάσεις και άτομα. Για παράδειγμα, μπορεί να περισυλλεγούν 40-50 και 5 ή 6 από αυτούς να υπάγονται σε αυτές τις κατηγορίες, να χρειάζονται τα χύτατα ιατρική περίθαλψη. Τι θα κάνουν τα κρατημέλη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αμέσως θα ε, συλλεγούν, θα περισυλλεγούν από ελικόπτερο και θα μεταφερθούν εκεί όπου χρειάζεται τα άτομα αυτά ώστε να έχουν την απαραίτητη φροντίδα. Τέτοιες ε, καταστάσεις υπάρχουν και πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε τα κράτη-μέλη να προσφέρουν την απαραίτητη αρρωγή. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι γιατί είναι τόσο πολλέ οι περιπτώσει, η περιπτωσιολογία τόσο ευρεία στο τι μπορεί να συμβεί που δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε όλα. Στο άρθρο 7, σωστά είπατε ότι υπάρχει ένα σφάλμα που πρέπει να διαγραφεί. Στο θέμα του αιτιολογημένη υποψία ή αιτιολογημένα υποψιάζονται, όχι. Και τελευταία ερώτηση στην επαφή με το κέντρο συντονισμού, θεωρείτε ότι το κέντρο συντονισμού θα ανταποκρίνεται σε ζητήματα, σε ερωτήματα, θα δίνει κατευθύνσεις, ενδεχομένως θα συντονίζει δηλαδή τις επιχειρήσεις διάσωσης. Και αν είναι κάτι λησμόνι, σε παρακαλώ υπερθυμίστε μου. Καλώς. Άλλα σχόλια υπάρχουν. Κύριε Κοέλιο, ο οποίος θα συντάξει κάποιο κείμενο εργασίας φαντάζομαι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όχι, θέλω να την Επιτροπή για τις απαντήσεις της. Και να υπογραμμίσω ότι πρέπει να εργαστούμε γρήγορα. Το θυμίζω σε όλους και τους συγκητές ε, που το επεσήμαναν οι ίδιοι ότι μπορούν να εργαστούν, πρέπει να το κάνουμε για να αντικατασταθεί η αποφάση του Συμβουλίου. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι και γρήγορα και να μην, να μην ξεχνάμε ότι όσο δεν έχει εγκριθεί ο κανονισμός μας ε, ε, ισχύει αυτή η αποφάση του Συμβουλίου. Αν δουλέψουμε λοιπόν γρήγορα μπορούμε να την ανατρέψουμε. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μέχρι εκεί για το συγκεκριμένο θέμα ήταν προσυζήτηση, μια προ Παρασκευή της συζήτηση. Το θέμα της Ουγγαρίας το επόμενο, που δεν είναι και ίσον σημασία, έχει προβλεφθεί για τις 11.45. Μισή ώρα μας περισσεύει. Ναι, και έχουμε λοιπόν προχωρήσει τόσο γρήγορα. Προτείνω διάλειμμα μισή ώρα και να ξαναρχίσουμε. Κυρία Κέλλαρ, εσείς. Ο Χουίς έρχεται. Πρόεδρε, σε ένα λεπτό θα είναι εδώ. Όχι, παρόλα αυτά, εγώ, εάν δεν έχετε αντίρρηση, κυρία Κέλλερ. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι έχουν προβλέψει ότι θα γίνει συνάντηση, η συζήτηση κάπου σε 11.45. Μισή ώρα για καφεδάκι στον ήλιο. Are we all set? Thank you. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Ευχαριστώ. Σημείο 9 λοιπόν. Όπως είχαμε προβλέψει. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις, ε, στην Ουγγαρία. «551 μόνο οι τροπολογίες στην έκθεση του κυρίου Ταβάρες. θα τον ακούσουμε και θα ακούσουμε στη συνέχεια τις συζητήσεις. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Όσο πιο σύντομα μπορώ. Έχουμε όντως 500 και τροπολογίες, πολλές οι επαναλήψεις. Πολλέ ναι, ναι, ναι. Πολλές οι επικαλύψεις. Ευχαριστώ όλους τους αδέλφου που κατέθεσαν τροπολογίες για τη συνεισφορά τους. Και βεβαίως θα προχωρήσουμε στην τακτική διαδικασία με τις συμβαστικές τροπολογίες, την σωμάτωση τροπολογιών στο νέο κείμενο, καταλόγους ε, ψηφοφοριών και το καθεξής. Η Ουγγρική κυβέρνηση επίσης απέστειλε τη συμβολή της. Κάποιες τροπολογίες οι οποίες θεωρώ πως μπορούν ε, κατά τρόπο σημαντικό να ε, ενημερώσουν, να επικαιροποιήσουν την έκθεση της ενσωμάτωσα. Αλλά πρέπει να πω ότι υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις ουγγρικής κυβέρνηση και κάποιες τοποθετήσεις και συμπληρωματικά σχόλια από την κοινωνία των πολιτών, πολύ πιο δεξοδικά από αυτά της Ουγγαρίας, της Ουγγρικής κυβέρνησης, σχόλια επί των σχολείων δηλαδή. Για το κομμάτι το εμπειρικό της εκθέσεως πρέπει να σας πω ότι έχει περάσει επιτυχώς την δοκιμασία των ε, τοποθετήσεων, των θέσεων τρίτων πλευρών. Και νομίζω ότι είναι ένα δοκιμασμένο πλέον κείμενο. Έχουμε λοιπόν ένα νέο πλαίσιο νομοθετικό, ένα νέο πεδίο νομοθετικό που αλλάζει, που άλλαξε και που αλλάζει ακόμη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσουν κάποιες τροπολογίες στη λεπτομέρειά τους. Πρόκειται για το νέο νόμο για την εθνική ασφάλεια. Από ό,τι γνωρίζω και θα ήθελα επισήμως από τη θέση αυτή να ζητήσω από την Ουγγρική κυβέρνηση μια επίσημη μετάφραση του νόμου περί εθνικής ασφαλείας. Προβλέπετε ότι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ε, ανώτατοι αξιωματικτούχοι, δημοσίοι, δηλαδή υπάλληλοι, δικαστικοί, ε, διπλωμάτες, ε, διοικητές ε, δημοσίων ε, φορέων ε, που Ε, ασχολούνται με θέματα ευαίσθητα, τα κτλ. μπορούν ή θα υπάγονται καλύτερα σε παρακολούθηση ε, και των συνδιαλέξεών τους και γενικά επιτήρηση τέτοιου τύπου για 30 μέρες το χρόνο και αντίστοιχα ξέρω ότι ο αναπληρωτής εισαγγελέα εξέφρασε ανησυχίες προς τον νόμο αυτό τον έχει ήδη εγκρίνει το Κοινοβούλιο αλλά όπως είπα, περιμένω την επίσημη μετάφραση. Διότι τίθενται ζητήματα και προστασίας του ιδιωτικού βίου και πρόσβασης της ε, κυβέρνησης σε στο έργο της δικαιοσύνης, η παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απόλυψη βεβαίως και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ε, εξασφαλίσουμε τις, τα ένδικα μέσα για την αποκατάσταση εκείνων που ενδεχομένως απελήθησαν άδικα. για τις ε, τροπολογίες. Υπάρχουν δύο ειδών τροπολογίες. Καταρχάς διευκρινήσεις και προσθήκες στην έκθεση. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα ορισμένες από αυτές. Διευκρινίζουν στους κάποια σημεία της εκθέσεως. Τις δέχομαι και εγώ σε έναν βαθμό τις διευκρινήσεις παραδείγματι η σταγματική διαδικασία μέσα στο κοινοβούλιο, όχι την ε, διαδικασία των διαβουλεύσεων που κράτησε περισσότερο χρόνο, αλλά η επεξεργασία του σχεδίου μέσα στο κοινοβούλιο κράτησε μόνο 30 μέρες, 35 μέρες, ε, Χωρί να έχει και μεγάλη σημασία τώρα το 30, το 35. Και μετά έχουμε και κάποιες διαγραφές από τις τροπολογίες. Και θα ήθελα οι συνάδελφοι να μου πούνε τη γνώμη του, να μου πούνε ποιο λόγο έχουν να υποβάλουν τις προτάσεις για διαγραφή. Διότι πρέπει να πω ότι μερικές φορές βλέπω να μην συνάδουν με τα όσα έχουμε μέχρι τώρα πράξει στην Επιτροπή μας αυτές οι διαγραφές. Στο στην αιτιολογική σκέψη π και όπου έχουμε αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το χάρτη κτλ. εκεί που αναφέρεται στα προήμια των συνθήκων και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που μνημονεύονται στο προήμιο τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Θρωτήριο του Καταστατικού του Συμβουλίου τη Ευρώπη από τη διάκριση των εξουσιών μεταξύ των θεσμών, θεμελιωμένων σε ένα εύρυθμο σύστημα αμοιβαίων ελέγχων και συμποροποιών και λαμβάνοντα υπόψη ότι στα βασικά χαρακτηριστικά ενό τέτοιου συστήματο προλαμβάνει το σεβασμό τη νομιμότητα μαζί με μια διαφανή, υπεύθυνη και δημοκρατική διεργασία εφαρμογή των νόμων, η ασφάλεια δικαίου, ένα στέρεο δίκαιο ε, σύστημα αντιπροσωπευτική δημοκρατία, σε ελεύθερε εκλογέ και στο σεβασμό των δικαιωμάτων τη και όλα αυτά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό ενοχλεί και θα πρέπει να απαλληφθεί. σε μια αναφορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά αποτελούν δίκαιο εσωτερικό και αυτονόητο. Ένα άλλο ζήτημα που είχαμε σε ένα άλλο σημείο στο 3 εκεί όπου εκφράζουμε τη λύπη μα για το ότι η διαργασία εκπόνηση και έγκριση του γρικού θεμελιώδου νόμου δεν είχε διαφάνεια, άνοιγμα στην προτιμότητα και σε τελική ανάλυση συνενετική βάση που θα μπορούσε κανεί να αναμένει από μια σύγχρονη δημοκρατική σταγματική διαργασία, πράγμα συνεπώ που αποδυνάμωσε την ομότητα του ίδιου του θεμελιώδου νόμου. Ε, αυτό υπήρχε και στα έγγραφα εργασία, ήταν ξεκάθαρο. Δεν, δεν συμμετέσχε η, η αντιπολίτευση του Κοινοβουλίου. Είναι δεδομένο δηλαδή. Και δεν καταλαβαίνω γιατί. Να τα συζητήσουμε. Είναι πραγματικά γεγονότα. Α τα συζητήσουμε. Ε, μια άλλη πρόταση για διαγραφή 5 ή 6 σελίδων από την έκθεση, ε, θα αφαιρούσε βέβαια την ουσία της εκθέσεως, ε, θα στερούσε από το κείμενο τον πυρήνα του. Και γι' αυτό, όπως είπα, έχω έρθει εδώ περισσότερο για να ακούσω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι, όσοι έχουν καταθέσει τροπολογίες, είμαι στη διάθεσή του για οποιαδήποτε συζήτηση ή διευκρίνηση. θα έλεγα να δούμε εάν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικέ τροπολογίε και μάλιστα να το κάνουμε σε δύο φάσει. Δηλαδή, θα έλεγα να βρούμε τι συμβαστικέ τροπολογίε για τα πιο εύκολα θέματα, τι δέκα πρώτε θα έλεγα, και μετά να συζητήσουμε αν έχουμε ένα περιθώριο για ακόμη περισσότερε. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση και των τροπολογιών. Να ακούσουμε του σκιώδει ηγητέ. Και εγώ σκιώδη είμαι. Αλλά α ακούσουμε πρώτα του άλλου συναδέλφου. Τον κύριο Έγκελ πρώτα από τις πολιτικές ομάδες, οι σκιώδεις Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα τα καταφέρουμε. Έχουμε όχι μόνο την έκθεση αλλά και ένα σημαντικό αριθμό τροπολογιών επιτάπητος. Και βλέπουμε ότι αντικατοπτρίζουν οι τροπολογίες αυτές τη σοβαρότητα και την ε, επικοδομητική στάση, την οποία οι περισσότεροι εξημών τουλάχιστον ακολουθήσαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, που όμως δεν μπορεί να αποκρύψει και διαφορές θεώρησης ενώπιστων συζητήσεων, θα, θα πω, διαπραγματεύσεων για περαιτέρω λύσεις και δυνατότητες. Για το θέμα αυτό λοιπόν της θεώρησης, χωρίς να θέλω να αποκρύψω και τη δική μου προσωπική θεώρηση στα πράγματα, θα πω τέξεις. Έχω καταθέσει και εγώ αρκετέ προτάσει τροπολογία που αναφέρει ο και θα εξηγήσω το γιατί. Καταρχάς, Ο χρόνος ήταν σχετικά σύντομος για την ε, κατάθεση τροπολογιών, ιδιαίτερος, ε, και δεν ήταν δυνατόν, όπως θα ήθελα, να βγάλω 50 παραγράφους για να ζητήσω μια πλήρη ε, αναδιατύπωση του, κινεύου, του κειμένου. Ούτε και μπορούσα βέβαια να κάνω λακτική έκθεση. Ένας από τους λόγους λοιπόν που κατέθεσα αυτές τις προτάσεις για διαγραφή ήταν για να επισημάνω ότι αυτό που υπόθηκε μπορεί να υποθεί, μπορεί να μην υποθεί, μπορεί να υποθεί με διαφορετικό τρόπο. Και να εξηγήσω τους λόγους που το πράττω αυτό. Γιατί θέλω να ζήσω από τον ε, συντάκτη ε, να επανεξετάσει της, ε, τη διατύπωσή του. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου ριζικά ζητώ τη διαγραφή, ξέρω ότι υπάρχουν εναλλακτικέ στη διατύπωση και όλες αυτές οι εναλλακτικέ διευκρινήσεις και όλα αυτά θα μπορούσαν να με ικανοποιήσουν, θα μπορούσα να τις δεχθώ. Άρα δεν χρειάζεται να παραμείνουν όλες τις τροπολογίες που προτείνουν διαγραφή από πλευρά μου. Αλλά θα απαντήσω απευθεία στον εισηγητή στο ερώτημα γιατί να διαγράψουμε κάτι το αυτονόητο. Και η απάντησή μου είναι ακριβώς αυτή. Επειδή είναι αυτονόητο. και όταν είναι αυτονόητο μπορεί να ε, δηλώνει κάτι, η καταγραφή του, που εγώ δεν θέλω να δηλωθεί. Ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να το θέλουν. Δηλαδή αν, πούμε, αν κάνουμε μια καταγραφή πλήρη των ε, στοιχείων που καταρτίζουν μια δημοκρατία, των χαρακτηριστικών μιας δημοκρατίας, βεβαίω δεν μπορώ να έχω αντίρρηση. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ε, ότι σε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οποίο κανεί δεν ισχυρίζεται ότι έχει εκπνεύσει η δημοκρατία πρέπει να υπενθυμίζουμε διαρκώς ότι πρέπει να είναι μια ορθώς λειτουργούσα δημοκρατία. Αυτό. Γι' αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε άλλες, ζητώ τη διαγραφή. Όχι γιατί δεν πιστεύω στις αξίες αυτές, αλλά γιατί ακριβώς πιστεύω στις αξίες αυτές και τις θεωρώ δεδομένες και δεν θεωρώ ότι πρέπει να τις επανακαταγράφουμε και να τις επαναφέρουμε στην συζήτηση που αφορά μια συγκεκριμένη χώρα και συγκεκριμένε συνθήκες που θα υποδήλωναν ενδεχομένω ότι έχει εγκαταλείψει τις δημοκρατικές διεργασίες η χώρα αυτή. Και επίσης θα ήθελα εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδα να εκφράσω την επιθυμία να επικεντρωθούμε στα πιο ουσιώδη στοιχεία και γι' αυτό οι, κάποιες άλλες προτάσεις τροπολογίας με διαγραφή και ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε εδώ με τη γενικότερη θεώρηση γιατί πολλά πράγματα είναι ζήτημα ερμηνείας. Πολλά πράγματα ερμηνεύονται κατά έναν τρόπο ή μπορούν να ερμηνευθούν κατά διαφορετικό τρόπο και επιτρέψτε μου να έχω την άποψή μου για την ερμηνεία αυτή, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν θεσμικά όργανα, υπάρχουν φορείς, οργανισμοί ανεξάρτητοι που έχουν ερμηνεύσει ε, κατά κάποιον τρόπο συγκεκριμένο τις ε, καταστάσεις, ενώ η Ουγγρική κυβέρνηση πάντοτε εκφράζει μια διαφορετική θέση και την... Ε, και την θέση της Ουγγρικής κυβέρνησης, η οποία εξηγεί, ερμηνεύει ποιες είναι οι ε, ποιος είναι ο σκοπός που εξυπηρετεί με την τροποποίηση, ποια είναι τα μελήματα που προσπαθεί να ε, προστατέψει. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία στα πράγματα ως εκ του, του οι τροπολογίες περί διαγραφής. Και ολοκληρώνω σε αυτήν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με το θέμα της θεώρησης στην έκθεση. Ξέρετε ότι ως κοιόδης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν θέλω να οδηγηθώ σε μια σαφή διαφωνία ή σύγκρουση. Ενδέχεται βεβαίως και το αποδέχομαι λόγω και πολιτικών προτιμήσεων, επιλογών, να μην φανούν τα πράγματα τόσο εύκολα όσο θα θέλαμε. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι είναι μια δυνατότητα η ευκαιρία αυτή και μπορεί να αποτελέσει μια δυνατότητα βλέπετε ότι έχω εμπιστοσύνη στον εισηγητή, να αποτελέσει ένα, μια ευκαιρία για προσδιορισμό μία θέσεως για το πώς συντάσσονται τα συντάγματα, ποια πρέπει να είναι η συνταγματική πρακτική, ποια πρέπει να είναι η συντακτική πρακτική, χωρίς να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο κράτος. Ε, υπάρχουν πράγματα στο οποίο έχει τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με διατεθειμένο να το δεχθώ και εγώ, ότι έχει ένα ρόλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Έχει ένα ρόλο να επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επιτέλεση του ρόλου αυτού δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τον κανένα. Αλλά μετά έρχονται οι πολιτικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις. Και για αυτές εγώ θα έλεγα ότι είναι προτιμότερο να υιοθετήσουμε μία στάση όπου θα προτείνουμε αντί να απειλούμε και θα καλούμε αντί να ζητούμε με έμφαση. Και θα πρότεινα πέραν τη συγκεκριμένη ευκαιρία που προσφέρεται με αυτή την ε, έκθεση να φτιάξουμε έναν, ε, μία βάση πάνω στην οποία θα στηριζόμαστε για περαιτέρω τοποθετήσεις, γιατί σε τελευταία ανάλυση πέραν των άρθρων αυτών του θεμελιώδους χάρτη κτλ. Δεν ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Τι σημαίνει προτείνουμε τρόπο σύνταξη συντάγματος. Αυτό πρέπει να το λύσουμε και εδώ καταλέγω, γιατί πρόκειται μια έκθεση για την Ουγγαρία, είναι μια έκθεση για την Ουγγαρία, μεν, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και ουχή λίγες, έχουμε επισημάνει ζητήματα που γεννούν ανησυχίες, τα οποία δεν τα έχουμε δει μόνο στην Ουγγαρία και θα ήταν ζήτημα που γεννεί, γεννά ανησυχία και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε μια ευρωπαϊκή καταγραφή και συναντήληψη του τι είναι η κοινή πρακτική. Αυτό έχει πολύ περισσότερο νόημα πιστεύω. Από το να ε, στιγματίζουμε μία συγκεκριμένη περίπτωση. Προσπαθώ πάντα να μην ε, το γυρνάω στη φιλοσοφία, αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση αναγκαστικά μας οδηγεί σε φιλοσοφικές επιλογές. Προσπαθώ επίσης και να μην μακρηγορώ, γι' αυτό σταματάω τώρα την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θέλω να σε εδώ στις λεπτομέρειες των τροπολογιών, γιατί ο συνάδελφο Ταβάρης και σχολίασε. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να τονίσω κάποια θέματα πολύ βασικά του δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε όταν συζητάμε για τροπολογίε, για συμβιβαστικέ διατάξει. ε, γενικά για την επεξεργασία αυτή τη έκθεση και θα πρέπει να συμβαίνουμε τον κύριο Αγγελίου όταν λέμε ότι αν θέλουμε να βλέπουμε να εφαρμόζουμε τρομερά δικαιώματα και δημοκρατία, κάτι το οποίο αφορά όλες μας τις τροπολογίες, τότε είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί κάτι ούτω ώστε να επικρίνουμε όλα τα κράτη-μέλη και γι' αυτό και ακριβώς αυτό το οποίο θέλω είναι να υπάρχει ένα πίνακα επιδόσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ώστε να μπορεί να γίνεται ο έλεγχος. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι συζητώντα για την Ουγγαρία, αυτό σημαίνει ότι δεν ε, ασχολούμαστε μόνο με ένα σημείο, ένα πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί ε, σημείο επίκρισης. Αλλά έχουμε μία σειρά ε, συζητήσεων, ένα σωρά ζητημάτων και αυτό γίνεται κάθε φορά που μιλάμε με εκπροσώπους της κυβέρνησης και δύο φορές είπαμε ότι μπορούμε, ε, ερχόμαστε σε μαζί του τέλος πάντων γιατί η συζήτηση ε, δεν είναι για το πώ θα γίνουν οι αλλαγέ. Το θέμα δεν είναι πώς εμείς βλέπουμε τα πράγματα ως ε, Ούγγροι, ως Ουγγρική κυβέρνηση, γιατί κάνουμε κάτι. Το ζήτημα είναι γιατί να τους επικρίνουμε κάθε φορά και πριν από λίγα χρόνια, ίσως το 2007, γιατί δεν είπαμε τίποτα, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί δεν ήμουν εδώ τότε. Πάντως, εφόσον ε, ισχύει το ότι έγιναν κάποια στραβά πριν μερικά χρόνια και κανεί δεν έκανε τίποτα, ε, εντάξει, αυτό ίσως είναι λάθος. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα, όταν σημαίνουμε κάποιο πρόβλημα, ότι δεν θα πρέπει να επικρίνουμε. Φυσικά και πρέπει. Και σε σχέση με την συνήθεια τη Λισαβόνα δεν είναι μόνο ε, δικαίωμα, είναι και υποχρέωσή μας να το συζητάμε. Επομένως νομίζω ότι υπάρχει κάτι το ειδικό για το τι γίνεται στην Ουγγαρία και θα πρέπει να τσεκάρουμε την ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα κρατημέλια. Αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να μπορέσουμε κάτι να, να, κάπου να καταλήξουμε ούτως ώστε με επιχειρήματα να μπορούμε να σταθμίσουμε όλες τις απόψεις. Και κοιτάξτε τι συζητήθηκε στις τελευταίες εβδομάδες, ε, πώς, πώς διαπιστώθηκε ότι επιβάλλεται να γίνουν κάποιες επικρίσεις, μα όταν ε, ε επικρίνεται πούμε, το Συμβούλιο, αυτό δεν είναι έργο κάποιων αριστερών γενικά, επομένως το θέμα δεν είναι να ζωρίσουμε την Ουγγαρία ή να πετάξουμε την Ουγγαρία έξω την Ένωση. Με μεγάλη μας χαρά επιστώνουμε ότι ανοίγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η να πεταξουμε την ουγγαρια εξω την ενωση με μεγαλη μα χαρα επιστωνουμε οτι ανοιγει στην ευρωπαικη ενωση η ουγγαρια Για, για, για, κοιτάξτε τι πέρασε στην ιστορία της αυτή η χώρα. Είναι πολύ θετικό το ότι τώρα ανήκει σε αυτή μας την κοινότητα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως έχουμε την υποχρέωση να παρακολουθούμε για, για το ότι τα πράγματα γίνονται σωστά, ότι εφαρμόζονται δικαιώματα κλπ γιατί υπάρχουν πάρα πολλά για τα οποία μπορεί κανείς να επικρίνει αλλά θα πρέπει βεβαίω να ελέγχονται όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε γι' αυτό σας λέω ελπίζω ότι θα αποφασίσουμε κάτι τελικά και θα αναβαθμίσουμε αυτές τις αξίες, ε, θα τους δώσουμε νόημα το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι το οποίο πάει παραπέρα. Γιατί θα πρέπει, αυτό το πρόβλημα παντού ότι τα θεμελιώδη μου είναι σημαντικά. Θέλουμε όλοι να προσέχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, αυτό, τελειώνω και τελειώνω, αυτό αν θέλουμε να ισχύει αλλού θα πρέπει πρώτα απ' να ισχύει και εδώ μέσα στο σπίτι μας. Αυτό το, για το οποίο επικρίνουν άλλους. Άρα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και για την Ουγγαρία και για όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να σας πενθυμίσω, λέει ο Πρόεδρος, ότι 12.30 θα πρέπει να ολοκληρώσουμε ω είναι τη συνεδριασή μα για σήμερα το πρωί. Πάντως βλέπω όλοι είναι και περισσότεροι ζητούν το λόγο όπως γίνεται συνήθως, οπότε παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι το 12.30 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Κύριε το με το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα είμαι σύντομη. Πρώτα πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταβάρες για τη δουλειά του, γιατί γνωρίζω πόσο δύσκολα ήταν ε, τα πράγματα και άλλωστε συνεχίζεται η δυσκολία και επίσης θα πρέπει να σας ε, πω σε όλους τους συναδέλφους από την Άλτε ότι θα πρέπει να, ισχύσει ε, το άρθρο 17 παράγραφος 1 της συνθήκης. Θα πρέπει επομένω να ισχύσει για τα κράτη-μέλη που δεν σέβονται όσο έχουν αποφασιστεί στην Κοπενχάγη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν δηλαδή τα μέσα να πιέσουμε τις χώρες να τηρήσουν τα, τα, τα υπεσχημένα, τα συμπεφωνημένα. Ε, δηλαδή πριν την ένταξη ε, είναι όλα καλά, αλλά και όταν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι θα πρέπει να αναλυθεί δράση, να αποδειχθεί πόσο σοβαρές είναι αυτές οι διατάξεις. Το άρθρο παράγραφος 1 θα πρέπει τώρα να το επικαλεστούμε. Και όποιος κάποιος ήδη ανέφερε, ίσως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πέραν της Ουγγαρίας για τις οποίες θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε αυτό το άρθρο. Τα κράτη-μέλη δεν είναι δυνατόν να μη σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα και να τη κλειτώνουν. Συνάδελφοι, εάν το 7.1 δεν χρησιμοποιηθεί τώρα για πρώτη φορά, ε πότε θα το χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί κάποιος να μου βρει ένα καλύτερο παράδειγμα εφαρμογή ή τώρα ή ποτέ. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αυτή τη συνταγματική τροπολογία αναλύεται, την ερμηνεύεται. Επίσης, ας κάτσουμε και σκεφτούμε κάτι το οποίο ένα από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ιδρύθηκε για να προστατεύσει τα δικαιώματα των κρατών μελών θα πρέπει πάντοτε να υπεραμείνετε των δικαιωμάτων των πολιτών. Επίσης, σας επισημαίνω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας για την τέταρτη συνταγματική τροπολογία. Πρόκειται για τρισέλιδο κείμενο. Θα πρέπει να μας προβληματίσει. Επίσης, θα ήθελα να σας παραθέσω τι λέει το συμπέρασμα στην τρίτη σελίδα. Η τέταρτη τροπολογία αφορά τα προβλήματα της δικαστικής εξουσίας, δηλαδή όσον αφορά την συνταγματική μεταρρύθμιση στην Ουγγαρία. Θέτει εν κινδύνο το Σύνταγμα και τις ε, του δικλείδες. Επίσης, την ε, εφαρμογή του κοινού νόμου όπως επιθυμεί η κοινωνική πλειοψηφία. Η τέταρτη τροπολογία θέλει να χειραγωγήσει για χάρη της πολιτικής το Σύνταγμα. Αυτό είναι δείγμα της κατάργησης της διάκρισης μεταξύ πολιτικής και συντάγματος. Θα πρέπει ή τώρα ή ποτέ να επικαλεστούμε να εφαρμόσουμε το άρθρο 7, παράγραφος 1. Θα σας δώσω το λόγο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε φτάσει στις 12 και 4. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια λίστα. Κύριε Άντς, δεν ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Μανχιστίν Γαρζά, της που είναι αρμόδια εκ μέρους της ε, ε, ομάδας μας να παρακολουθεί το θέμα αυτό. Θα ήθελα να παρουσιάσω την έκθεσή της, ε, την δική της τοποθέτηση στην έκθεση. Καταρχάς, υποστηρίζουμε απολύτως την έκθεση. Είναι μια από τις πιο σημαντικές εκθέσεις πρωτοβουλία της θητείας μας. Τέτοια σημασία αποδίδουμε στην έκθεση αυτή. Και γι' αυτό για το αν θα πρέπει να γίνει μια επαλήθευση της στήριξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τα κράτη-μέλη, ε, η απάντηση για μας είναι ναι. Ε, στα υποψήφια κράτη-μέλη γίνεται αυτή η επαλήθευση. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και στα κράτη-μέλη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφορά μόνο την Ουγγαρία η διαπίστωση των σφαλμάτων ή των προβλημάτων προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και πολλά άλλα κράτη-μέλη. Αλλά πρέπει όταν διαπιστώνονται προβλήματα να το πράττουμε και δεν θα πρέπει να παίζει ρόλο το αν τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται και σε άλλα κρατη κράτη-μέλη ή άλλα προβλήματα. Άρα χρειάζεται μια επαλήθευση, ένα check-up τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν ε, υπάρχει η αρχή απαράβατη ότι λειτουργεί μια δημοκρατία χωρίς προβλήματα στα κράτη-μέλη και ότι η Ουγγαρία δεν έχει κανένα πρόβλημα δημοκρατίας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μπορεί να προκύψουν ζητήματα και όντω ε, προκύπτουν και γι' αυτό είναι και ενσωματωμένα στην έκθεση. Όσον αφορά τι δικέ μα τροπολογίε, πολύ σημαντικέ για μα και θα θέλαμε να στήσουμε από τον ε, εισηγητή να τι λάβει υπόψη, πρόκειται για την τροπολογία 25 καταρχά Όταν μιλούμε λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να, μιλούμε, να αναφερόμαστε μόνο σε πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητέ φίλε, τα βάρε αν θέλει να το κοιτάξει άλλη μια φορά, γιατί και άλλα πρόσωπα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανεξαρτήτω τη ηθαγένειά του. Ανεξαρτήτω του αν είναι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεξαρτήτω τη ε, θρησκευτική του ε, πεποίθηση ή άλλων κριτηρίων. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Άλλο θέμα στην τροπολογία 76 που επίσης είναι σημαντικά για, σημαντική για μας, διότι επισημαίνεται με την τροπολογία αυτή ότι ε, η διαδικασία δεν τηρήθηκε σωστά στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Δεν ελήφθη υπόψη η τοποθέτηση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, αλλά μόνο της φίδες και του συνασπισμού του κυβερνητικού. Επίσης, το θέμα των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκπομπών ε, είναι ένα θέμα που επισημαίνεται με τροπολογία 495. Είναι πολύ σημαντικό ε, το πώς επηρεάστηκαν ή πώς λειτουργήσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διαδικασία αυτή. Και εν τέλει μιλάμε για τις διαδικασίες υπαραβάσης των συνθήκων και νομίζω ότι θα πρέπει το ζήτημα αυτό να το ε, χειριστούμε πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό στην τροπολογία 378 επισημαίνουμε το σχετικό αίτημα. Εν γέννη πάντως δεν θέλω να πω ότι κρίνουμε θετικά τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο λόγω του άρθρου 7, και όχι μόνο μια παραπομπή δηλαδή στο άρθρο 7, γιατί θεωρούμε ότι δεν αρκεί, θα θέλαμε να θεσπίζεται και προκαταβολικά η παρακολούθηση της αυστηρής στήρησης των αρχών, των θεμελιωδών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κάλλα, προσέξτε. Δεν έχουμε ώρα. Δεν πρέπει να ξεπεράσουμε το χρονικό όριο. Δεν, δεν θα τα καταφέρουμε αλλιώ. Μην το ξεχνάτε. Ναι, ναι, δεν θα είμαι σύντομη, λέει η κυρία Γκάλ. Ανέφερε ο συγκεκριτή ότι έχουμε επαλείψει ένα σωρό παραγράφου. Ναι, είναι αλήθεια ότι ζητήσαμε να επαληθούν όλε αυτέ τι παράγραφοι, εκείνε που αφορούν ερμηνεία. Επίση, αναφέρεται το άρθρο 2. Εμεί μελετήσαμε το άρθρο 2. Ε, τώρα περιέχει την ουσία του άρθρου 2, αλλά όχι την ερμηνεία. Επίσης ζητήσαμε την απάλληψη όλων εκείνων των σημείων που δεν αφορούν αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής, που είναι θέματα εθνικής κυβέρνησης. Θέματα που ποτέ δεν ετέθησαν εδώ. Δεν ξέρω. Θα σχολιώσασταν με θέματα κυβέρνησης της δικής σας χώρας. Τι θα λέγανε οι εθνικοί βουλευτές των χωρών σας. Ζητήσαμε να παληφθούν λοιπόν όλα τα σημεία στα οποία η Επιτροπή μα τοποθετείται και εκφράζεται ως δικαστήριο. Ε, βέβαια δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι κύριε Βίξτρομ, διατυπώνεται εδώ πέρα η άποψη ότι παραβίαση των δικαιωμάτων, αλλά δεν αποδεικνύεται. Απλώς κάνουμε μια γενικόλογη συζήτηση. Οπότε ας κρίνουν για το τι έγινε τα δικαστήρια. Επίσης για τα υπόλοιπα σχόλια θέλουμε να πούμε ότι έχουν γίνει διάφορα λάθη, πολλά λάθη και έχει διαστρεβλωθεί η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχουμε προτείνει κάποιες τροπολογίες και αφορούν την ερμηνεία του πώς εσείς βλέπετε τους νόμους, δικαστικές αποφάσεις, ε, διάφορα ζητήματα που είναι υποκειμενικά. Και θα μπορούσε κανείς αντί για αυτό το κομμάτι ας πούμε, της δικαστικής να βάλει ένα άλλο και να αλλάξει τελείως η εικόνα. Επομένως όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Επίσης, έχουμε τροπολογίες σε όλα τα σημεία στα οποία προκύπτει ότι κανείς δεν έχει επικρίνει άλλο κράτος μέλος για τα ίδια πράγματα. Ξαφνικά όμως όλα αυτά που ήταν παραδεκτά κατέστησαν απαράδεκτα και αφόρητα στο δίκτυο της Ουγγαρίας. Τώρα για τη συνάδελφο που έλεγε τι, τι, τι έγινε πριν και δεν υπήρχε καμία επίκριση. Ε, ακριβώς αυτό αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι πολιτικού χαρακτήρα. Αν είχαμε σωσιαστική κυβέρνηση τώρα στην Ουγγαρία, όλα αυτά δεν θα πίεζαν κανέναν γιατί όλα αυτά γινόταν από την αρχή του, του 90 και κανένα τώρα δεν θα είχε ε, ε πειράχτη επομένω. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτές οι επικρίσεις είναι διομετρική δύο σταθμά, ότι είναι έντονα πολιτικοποιημένου, πολιτικού χαρακτήρα. Τέλος πάντων, εδώ βάζω τελεία. Κύριε Βάιντεν, Χόλτσον και εσείς παρακαλώ να είστε σύντομος. Τρία σημεία ουσιαστικά. Έχει γίνει συζήτηση στην Κοπενχάγη ε, για τα κριτήρια της Κοπεχάγης, αν θα πρέπει να τα περιλάβουμε ή όχι. Ε, ούτως ή άλλως όταν γίνεται κανείς μέλος επαληθεύονται και μετά λέτε δεν πρέπει να ε, Αυτό δεν θα το συστήσω. Δύο παράγοντες όμως θα ήθελα να επισημάνω. Πρώτον, ο παράγον χρόνος. Έχουμε μια απόφαση του Φεβρουαρίου 2012. Έχει πέρασει ένας χρόνος. Ε, ακόμα δεν, δεν είχαν εκριθεί τα θέματα. Εν ε, παρισφρίουν νέε εξελίξεις και άρα πρέπει να καταλήξουμε σε μια απόφαση για να είμαστε θέση να διατυπώσουμε μια θέση, μια τοποθέτηση με σημασία, ίσως κάποια πράγματα να μην είχαν υποθεί εάν είχαμε καταλήξει νωρίτερα σε μια απόφαση. Και δεύτερον, να και πρόγραμμα για τον οικοκράτος έχω παρατηρήσει ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε αντίστοιχες ε, καταστάσεις με κυρώσεις οι οποίες ήταν εσφαλμένες, εσφαλμένη επιλογή, λάθος ε, τοποθέτηση, αντιπαραγωγικές και τελικά οδηγούν και σε μια ε, ανάπτυξη ε, νοοτροπίας ότι υπάρχουν εξωτερικοί εχθροί και σε μια αναδίπλωση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποφύγουμε γιατί ούτε την Ουγγαρία βοηθάει ούτε εμάς. Εδώ δέχω την εντύπωση ότι σε αυτό το θέμα όλο και περισσότερο επικεντρωνόμαστε και θα αναφέρω δύο θέματα της τροπολογίας ε, της, τροπολογίας της κυρίας Γκάλ ότι αντίστοιχα και στην Αυστρία είχαμε τέτοια ζητήματα. Μα ακριβώς αυτό είναι που επικρίνει ο κόσμος στην χώρα μας, ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, γιατί με τέτοια συζήτηση μας οδηγεί ακριβώς εκεί που δεν θέλουμε να πάμε, ότι δηλαδή ε, μπορεί αυτή η κακή πρακτική, κάτι το λάθος μπορεί να επεκταθεί και να διαδοθεί και να επιμολύνει τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν εκεί ακριβώς όπου υπάρχουν, όπου υπάρχουν πλειοψηφίες των δύο τρίτων και έχουμε και αντίστοιχες προτάσεις όχι μόνο στις στα αλλά και στις Ρουμανίες έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτές οι πλειοψηφικές, οι ειδικές πλειοψηφίες των δύο τρίτων έχουν βαρύτητα αντίστοιχη με ενός συνταγματικού Δικαστηρίο και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Η έκθεση δεν πρέπει να αφορά την Ουγγαρία πρέπει να μας αφορά όλους και δεν αποκλείω το δικό μου το κράτος από αυτό το όλους. Η συζήτηση πρέπει να γίνει, πρέπει να διδαχθούμε από αυτήν, αλλά δεν πρέπει και να διώξουμε ένα κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σύντομο και σαφές το μήνυμά σας. Τώρα έχω διάφορα μέλη του ΕΛΚ. Ε, για να τελειώσουμε. Κυρία Γιάροκα, σας ευχαριστώ πολύ για τις διαγραφές, γιατί έχουμε ζητήσει διαγραφές με τις τροπολογίες μας, γιατί υπάρχουν ε, όπως στο ενατολογικό και η σκέψη ε ή α, όπου υπάρχουν ε, λογικές, ε, λογικά σφάλματα. Επίσης ζητήσαμε διαγραφές στις μονόπλευρες αλήθειες, όπως στο ε, B και AC, οι, εκτιμο, οι σκέψεις λένε για τον θεμελιώδη νόμο, σαν να μην ε, ήταν αναπόσπαστο τμήμα του συντάγματος. Επίσης, νομικά σφάλματα που θα θέλαμε να διαγράψουμε από τα κείμενα, στην παράγραφο 12, που λέει ας πούμε η συνταγματική δικαιοδοσία σε σχέση με τον κεντρικό προπολογισμό θα, αποδι... θα εμποδίσει την αποδυνάμωση των ε, θεσμικών οργάνων και των εγγυήσεων. Νέες τροπολογίες ε, τώρα που έχουμε υποβάλει ε, είναι, αφορούν παραπλανητικές παραβλέψεις ή παραλήψεις. Εδώ λέει ότι γίνονται περισσότερα εγκλήματα μίσους. και ρατσισμού πιο συστηματικά υπ' αυτή την κυβέρνηση. Το να βάλουμε αυτή την παράγραφο στο τμήμα αξιολόγηση των μέτρων της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη ο σύνδεση με την εμπειρική κυβέρνηση, το απορρίπτω κάθετα και ρώτησα από τον εισηγητή, ζήτησα μάλλον από τον να δει μια ματιά να, στους νόμους που αφορούν την απαγόρευση των ακραίων ε, ομάδων ή την επινικοποίηση του λοκαυτώματος και τα λοιπά. Και εκεί η εικόνα είναι πολύ προκατηλημένη. Η Ουγγαρία είναι μοναδική, όχι μόνο διότι έχει βάλει τις στοχότερες μειονότητες ε, στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης, αλλά επίσης, για παράδειγμα, το ντοσχέ Ρώμα είναι στην υψηλή προτεραιότητα όλων των κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Έχουμε επίσης γύρω τραπέζες κατά των διακρίσεων. Είναι η μόνη χώρα η Ουγγαρία όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα κοινωτικά κονδύλια ε, ή στην χρηματοδότηση εφόσον ισχύσει το, όντως το πρόγραμμα ίσων ευκαιριών. Και είναι η μόνη χώρα στην χρηματοδοτηση εφοσον ισχυσει το οντως το προγραμμα των ευκαιριων και ειναι η μονη χωρα στην ουγγαρια που ισχύει σοβαρή νομική συνεργασία με τους πραγματικούς εκλογμένους εκπροσώπους των Ρώμα. Οπότε υπάρχουν τουλάχιστον αποτελέσματα. Είμαι στεκατά των τμήματων της έκθεσης όπου ε, αναφέρονται διάφορες αυθαίρετε απαιτήσει που δεν στηρίζονται από την κοινοτική νομοθεσία. Ευχαριστώ κυρία Ματιέ. Κοιτάξτε, του χρόνου έχουμε ευρωεκλογέ. Φαντάζομαι πω όλοι κοιτάτε τι δημοσκοπήσει. Για δείτε λίγο τι γίνεται με την ακροδεξιά που ε, παίρνει πάνω τη σε όλη την Ένωση και θα ήθελα να βρούμε συμβιβαστικές σε αυτή την έκθεση γιατί δεν θα ήθελα ε, να επικρατήσει ένας ευρωσκεπτικισμός και να οξυνθεί τόσο στην Ουγγαρία όσο και στην Ένωση. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα όσα έγιναν το 2010 με το ψήφισμα που είχαμε για τους Ρώμα. Ε, δεν έχει νόημα η ουσία, αλλά υπήρξε μια απόρριψη στο πλαίσιο των Γάλλων που είπαν ότι αρκεί, ε, φτάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας λέει και τι θα κάνουμε ε, μέσα στο κράτος μέλος μας. Αυτό ένα προήμιο, να προσέχετε λοιπόν. Προσοχή, προσοχή. Και τώρα είπα, υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία βρίσκουμε, εδώ τα βλέπω στα γαλλικά, τα βλέπουμε και εμείς στη Γαλλία, για παράδειγμα, για την δημοσιότητα των πολιτικών, για την αλλαγή τη εκλογική διαδικασία, Για παράδειγμα, με τις εκλογές που έχουμε του χρόνου, η κυβέρνηση τροποποιεί τους κανόνες των εκλογών. Και εμείς το έχουμε κάνει. Δεν, λέω, δεν επικρίνω τι είναι η σοσιαλιστική κυβέρνηση και το EMP το έκανε πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις. Κανένας δεν είπε τίποτα στη ΛΥΜΠΕ. Είναι μια συνήθεια στη Γαλλία ένα χρόνο πριν τις εκλογές να τροποποιείται να τρυποποιούνται οι περιφέρειε εκλογικέ. και κανένα στη Λίμπε δεν εκπλήσεται γι' αυτό. Αντίθετα όμω, επειδή είναι στην Ουγγαρία τώρα μα εντυπωσιάζει για την ε, δημοσιότητα των πολιτικών, ναι. Όντω κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι συνάδελφοι παρενέβησαν και πιστεύω πω ε, τονίζουμε υπερβολικά την Ουγγαρία και δεν είναι πολύ φρόνιμο αυτό. Η, του, η παρέμβαση του σοσιαλιστή αυστριακού συναδέλφου είναι πολύ φρόνιμη είχε χρησιμοποιήσει το σωστό τόνο και θυμηθείτε τι έγινε πριν από λίγα χρόνια με την άφηξη του Χάιντερ στον κυβερνητικό συνασπισμό. Φανταστείτε λίγο τον αυστριακό λαό, τι έζησε τότε. Ίσως λοιπόν θα πρέπει κάπως να ρίξουμε τους τόνους και να μειώσουμε την πίεση. Όσον αφορά το ΕΛΚ, θα φαντάζεστε κυρία Βίξτρομ ότι προφανώς η εφαρμογή του 7 δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Και φυσικά θα το καταψηφίσουμε. Όπως και αρκετοί από εσά ήμουν στο ημικύκλιο όταν ο, παρενέβη ο Πρωθυπουργός Ορμπάν και είπε ότι θα κάνει κάποιες αλλαγές, όλες αυτές που επιθυμούσε δηλαδή το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και ελπίζω πως θα τηρήσει την υπόσχεσή του, τουλάχιστον εγώ τον εμπιστεύομαι για τα όσα έχει ήδη κάνει, έχει ήδη κάνει κάποιες αλλαγές και τώρα περιμένουμε τις επόμενες. Ευχαριστούμε κύριε Ματιώτη. Κοιτάξτε, παρακαλώ σύντομα. Σύντομα μας τέλειωσε ο χρόνος. Και πρέπει να πάρω και εγώ το λόγο. Είμαι σκιώδη σε αυτή την έκθεση. Θα, θα, δεν θα ακριβωρήσω, αλλά ε, κοιτάξτε, εγώ θα είμαι πολύ σύντομα. Βρίσκω αυτή τη συζήτηση πολύ κουραστική και θεωρώ πως είναι μια χαμένη ευκαιρία. Ναι, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι είναι άδικο, πως έχουμε επικρίνει ότι δεν έχουμε επικρίνει άλλες κυβερνήσεις και τα λοιπά, αυτοί που λένε ότι αυτό προκαλεί αρνητική αντίδραση στη χώρα και τα όλα αυτά είναι αλήθεια, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να συζητήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην πραγματικότητα και όχι μόνο σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε αρκετά. Η κυρία Ματιέ λέει πως είναι ατυχές ότι απομονώνουμε και καταδεικνύουμε μία μόνο χώρα. Όταν ξεκίνησε όμως αυτή η υπόθεση, εγώ προσωπικά πρότεινα να γίνει μια έκθεση γιατί τότε ήταν το θέμα η ελευθεροτυπία, να γίνεται ετήσια έκθεση από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για όλα τα κρατημέλια. Ακριβώς για να αποφύγουμε αυτό που είπατε. Αλλά το απορρίψατε. Το απόρριψε το ΕΛΚ. Εσείς χάσατε την ευκαιρία τότε. να διευρύνετε την ε, ε, έμφαση που δίνεται από για μια χώρα σε όλες τις χώρες. Ε, και πιστεύω πως θα, είμαστε, θα είναι και λίγο πιο ανοιχτή η χώρα. Υπάρχει αρνητική αντίδραση, ναι, και το καταλαβαίνω ποια είναι η ψυχολογία. Ακόμα και αν δεν είμαι Αυστριακή, μπορώ να φανταστώ Όμως αν ταυτόχρονα σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να συζητάμε προβλήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, προβλήματα με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία που συμβαίνουν στα κράτη-μέλη, ε, τότε τι κάνουμε εδώ. Ε, Και φυσικά είναι δύσκολο και πονάει. Αλλά δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση Γιατί ας πούμε αν παραβιάζονταν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ε, φυσικά θα το θεωρούσαμε φυσικό να, επικρίνουμε το κράτος μέλος. Ενώ τώρα επειδή είναι θεμελιώδη δικαιώματα είναι ταμπού το θέμα. Είναι μεγάλο τεστ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Πρόεδρε είναι τελευταία μου παρατήρηση και είναι σημαντικό το θέμα. Εγώ Πιστεύω απόλυτα στην ακαιρεότητα όλων των συναδέλφων συμπεριλαμβανομένων των Ουγγρινών, των Ούγγρων και της ε, συμπαθεστά της συναδέλφου κάθε δίπλα μου. Έχω βαρεθεί όλους αυτούς τους χειρισμού που απευθύνονται προς τα κέντρο αριστερά κόμματα που λένε ότι όλα αυτά είναι ε, πολιτικής φύσης, λες και είναι καμιά συνωμοσία. Μα δείτε λίγο την κυβέρνηση ε, ΕΛΚ. Είναι κάποιοι, είναι αρκετοί εκεί και δεν είναι και πολύ καλοί για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πραγματικά δυσαρεστούμε ε, ε, όταν ε, κανείς αμφισβητεί την ακαιρεότητά μου. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο κομματικό. Και θα πρέπει να μην κάνουμε τέτοια σχόλια μεταξύ μας. Ναι, ναι, θα είμαι σύντομη γιατί πρέπει να προλάβω το αεροπλάνο. Δύο φράσεις. Διαβάστε την αναφορά της, της για την πολιτική, του για τους Ρωμά. Ε, Βερονίκη, ένα ε, πραγματικό περιστατικό. Δεν είμαι αντισημίτης ή ε, αντιευρωπαία ή αντιρωμά. Το, τελικά ε, η κυβέρνηση το θέμα είναι τι κάνει. Είχαμε δημοσιογράφους που παρασυμφορήθηκαν οι οποίοι ήταν φανατικά αντισημίτες και αντιρωμά. Είχαμε και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον ίδιο. Ο οποίος επίσης ήταν κοντά σε κάποιον ο οποίος ήταν επίσης αντιεβραίος αντισημίτης. Ένα ολόκληρο κατάλογο με τέτοια γεγονότα θα μπορούσα να σας πω, τέτοια στοιχεία. Επομένως, να, να ποια είναι τα δημιουργία δύο σταθμά. Δεν είναι το πρόσωπο που δείχνουν προς τα έξω και το δείχνουν τα μέσα. Κύριε Ταβάρες, όπως σας είπα είμαι ο ίδιος ε, σχεδοσυγητής αλλά εγώ δεν θα ε, λάβω το λόγο παρά μόνο για να σας πω δύο φράσεις. Πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο των σχεδόν γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει επομένω να βοηθήσουν και του να υπάρχει ισορροπία μεταξύ και να έχουμε κάποιε τροπολογίε που φυσικά είναι πάρα πολλέ. Περίπου 500. Και επίση υπάρχουν και αντιφατικέ. Ε, μεταξύ τους. Άρα θα πρέπει να βρεθεί η ισορροπία. Επίσης, σας είπα ότι η πολιτική μου ομάδα ανησυχεί όσον αφορά το σημερινό σύστημα, το δικαίωμα ε, κλείνει και κλαίγεστε και επίσης για το ότι φημώνεται κατά κάποιο τρόπο το στεγνωτικό δικαστήριο γιατί ακριβώς αποφάνθηκε σε σχέση με τις ε, τροπολογίες αυτές ή τις τροποποίησεις του δράγματος τέλο πάντων που ήθελε η πλειοψηφία και κυρίως ε, είναι και το θέμα της δικαιοσύνης και επίσης είχαμε και παρεμβάσει τη δικαιοσύνη κόντρα σε όσα έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Επιτροπή της Βενετίας. Ναι. Επίσης, σε όλη την Ευρώπη χρειάζονται ειδικέ πλειοψηφίε ούτω ώστε να αναθεωρηθεί ένα σύνταγμα. Δύο τρίτα στα περισσότερα συντάγματα. Γίνεται όμως γρήγορα, γίνεται συχνά. Οπότε με, με κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες επιβάλλονται κάποιες αλλαγές, αλλαγές που εξυπηρετούν πολιτικά. Και άρα σκεφτείτε. Ότι κατά αυτόν τον τρόπο χάνεται η ακρίβεια με την οποία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρεί τις υποχρεώσεις της. Να περιφρουρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το επιτάσσει η συνήθεια της αγώνας. Και άλλωστε το είπε και η κυρία Μπέναβα στην έκθεσή της και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη. Κάθε φορά που έχουμε μία πάρα πολύ σημαντική τροποποίηση συντάγματο που έρχεται αμέσω μετά από μία προηγούμενη, τότε θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος του κατά πόσο αυτά συνάδουν προς τα όσα συμβαίνουν στην Κοπενχάγη. Τα βάρε έχετε το λόγο. Ναι, θα είμαι σύντομο. Και βέβαια συνάδελφοι καταλαβαίνετε ότι μπορώ να απαντήσω σε όλους. Πρώτα πρώτα Να σου πω συνάδελφε, τι γίνεται με το πόσο κανείς μπορεί να το δει φιλοσοφικά. Υπάρχει και σχετικό της βέβαια που ανέκυψε σε όλη τη διαδρομή αυτή της έκθεσης. Τι θα πει η δημοκρατία, τι θα πει η κράτος δικαίου. Ε, αυτό είναι ε, υπερβολικά ε, σχετικιστικό. Να μην καταλήγω να είμαστε μηδενιστές, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Υπάρχουν κάποια πράγματα αυτονόητα. Κράτο δικαίου, δημοκρατία, δικαιώματα και αυτά είναι τα θεμέλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη μεριά όμω. Ε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε οποιαδήποτε ερμηνεία για το τι σημαίνουν ε, ε, θεμελιώδεις αξίες και αυτά. Ε, τότε, πια δεν είναι κανείς σχετικιστής, είναι μηδενιστής. Τώρα για τις ε, τροποποίησεις του συντάγματος, άκουσα τι είπε η κυρία Γκάλ, προσπάθησε να μην έχει πολύ υπογείμενο χαρακτήρα η έκθεση και εγώ επίσης έχω κάποιες τροπολογίες στο δικό μου το κείμενο και έχουμε και κάποιες ε, συμβαστικές τροπολογίες οπότε με όλα αυτά θα, σταμα... με όλα αυτά θα είναι όσο είναι πιο λίγο υποκειμενικό το κείμενο. Αλλά με κάποιες ερμηνείες μην φτάσουμε να καταστρέψουμε την έκθεση ή πάλι να ε, παραπέμπουμε σε άλλες χώρες. Υπάρχει τώρα επίσης και ο κίνδυνος των δύο δύο σταθμών. Ας πούμε, κάποιοι ανέφεραν την Αυστρία. Στην Αυστρία δεν εφαρμόστηκε κανείς νόμος, δεν εφαρμόστηκε κάτι, γιατί πρόκειτο για περίοδο πριν της συνδίκης της Λισαβόνας. Γιατί η συνδίκη της Λισαβόνας έφερε την αλλαγή στην αρχιτεκτονική του δικαίου ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και έτσι άλλαξε επομένως η κατάσταση. Το είπε και η κυρία Γκάλ στην έκθεσή της το 2010. Ε, θυμάμαι, τότε οι δράσεις ήταν ε, πάρα πολύ έντονες. Τώρα έχουμε πάνω από 500 σχετικούς νόμους. 49 ευξημένες ισχύω. Κυρία Γιαρόκα, ε, είπατε για αυτές τις ιδεολογίες ε, παραγράφους, α, β και εκεί λέμε ότι το Σύνταγμα της Ουγγαρίας θεσπίζει κάποιους νόμου ευξημένης ισχύω για 26-27 ζητήματα. Αυτό είναι γεγονός. Και συνέδευτο με όλα όσα βεβαιώνει η κυβέρνηση. Κάτι σε άλλες χώρες καλύπτονται περισσότερα σημεία. Εντάξει. Εντάξει, ισχύει αυτό. Αλλά όμως μέσα σε 1,5 χρόνο θεσπίστηκαν αυτοί οι 49 νόμοι στην Ουγγαρία. Περισσότεροι από αυτούς πέρασαν χωρίς συνεργασία της αντιπολίτευσης. Δεν το λέμε όμως αυτό. Αυτό είναι πραγματικό περιστατικό. Θέλετε να το σβήσουμε από την έκθεση. Ε, τότε τι θα μείνει. Το ίδιο ισχύει και για την λογική παράγραφο ε ή που η οποία παραπέμπει στο άρθρο 6 της Συνδίκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης λέει για τα συντάγματα Μελλον λέει για την προσχώρηση στην Σύμβαση Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων. Να, ένα από τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Κυρία Βίξεν, για το άρθρο 7, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, μας ανέφερε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας. Εγώ περιμένω ακόμη το επίσημο κείμενο, γιατί το μόνο κείμενο που έχουμε είναι ό,τι δημοσιεύθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται βέβαια για θέμα ευρύτερο τη εκθεσή μου, γιατί αναφέρεται σε επίθεση κατά του συντάγματο, κατά του συνταγματικού δικαστηρίου και ότι αυτό γίνεται εκ Αυτά όλα δεν τα λέω στην έκθεση, περιμένω το επίσημο κείμενο. όμω είναι αλήθεια και αυτό είναι επιλογή του ε, συντάκτη σα να μην βιαστούμε να εφαρμόσουμε το άρθρο 7. Γιατί έχουμε και άλλα προσωρινά μέσα όπως είπαν και οι συνάδελφοι του ΕΛΚ, για κάποιο είδους πάγια συνεχή εποπτεία. Πολλές φορές διαφωνούμε την κυρία Μέρκελ, αλλά εν προκειμένου συμφωνώ. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είπε πρόσφατα ότι θέλει κάποιο είδους ε, ενδιάμεσα μέτρα. Και γι' αυτό απευθύνθηκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κλείνω, τελειώνω, τελειώνω και είχαμε και την επιστολή των τεσσάρων πρωθυπουργών στη Γερμανία, κατοχώρηση κλπ. Για να απευθυνθούν στην Επιτροπή και να δούμε τι μπορεί να γίνει βάσει του Άρθρο 2. Και τι μπορεί να γίνει. Δεν έχουμε κάποιο θέμα που αφορά το άρθρο 2. Για την κυρία Ματιά τώρα. Είναι αλήθεια ότι σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να αλλάξει ο εκλογικό νόμος ένα χρόνο πριν τι εκλογέ. Και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνει υπόψη όταν έχουμε αυτούς τους πίνακε των επιδόσεων που προτείνει η κυρία Ρέντινγκ. Αλλά τέτοια πράγματα ακριβώ όπω εδώ για τα μέσα ενημέρωση, για τη δικαιοσύνη, τέτοιο, τέτοιο άλλο παράδειγμα δεν έχουμε. Μετά έχουμε την τέταρτη τροπολογία, τέταρτη τροποποίηση. Έχουμε το θέμα της ε, αναπομπής των ε, υποθέσεων από δικαστήριο σε δικαστήριο. Έχουμε το νέο νόμο για την κριτική ασφάλεια. Περιμένουμε την ε, μετάφραση τον άλλο για τον ιδιωτικό βίο, για την διάκριση των εξουσιών. σα ευχαριστώ όλου για τι τροπολογίε σα και περιμένω τη συζήτηση για τι συμβατικές τροπολογίες. Ευχαριστούμε εισηγητά, ευχαριστούμε όλου όσου έλαβαν το λόγο, παρακολουθούμε την εξέλιξη και θα συνεχίσουμε τη δουλειά σε αυτό το σημαντικό θέμα και θα κάνουμε έκτακτη συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Στις 7 ε, η ώρα, στις 10 του μηνός να συμφωνήσουμε για αυτό το δέσμη μέτρο για το Σέγγεν και το, το άσυλο και θα έχουμε και τη μάλιστα να μας πει για τη Ρωσία. Γεια σας, τα λέμε δεύτερο.